So, meine vereinzelten äh, Damen und Herren, oh, jetzt ist die Berichterstattung. Nein. Ladies and gentlemen. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε. The, uh, ladies and gentlemen who are here. Καλώ ήρθατε όσοι ήρθατε, εν πάση περιπτώσει. Αλλάξαμε την ημερήσια διάταξη. Και συζητάμε τώρα κάποια δήματα πολιτικής ουσίας. Θα είχαμε κανονικά την συζήτηση με τον ε, κύριο Ταγιάννη, ο οποίος όμως ακύρωσε αυτό το βράδυ, τελευταία στιγμή, δεν μπορώ, δεν ξέρω γιατί. Δεν ήταν κάτι το επίγον και πολιτικό, ό,τι και αν είναι αυτό. Εγώ, εν πάση περιπτώσει, θα το απευθύνω μια επιστολή εξ ονόματος της Επιτροπής, αν δεν έχετε αντιρρήσεις, για το ότι δεν είναι σωστό αυτό. Ναι, εμείς ε, προγραμματίζουμε, προσπαθούμε να βρούμε χρόνο που να βολεύει όλους και τώρα τελευταία στιγμή ε, μας προκαλεί και προβλήματα αυτό. Με πάση περιπτώσει τα σημεία 13 και 14 ήρθαν πρώτα πρώτα στην ημερήσια διάταξη. Οπότε θα ήθελα να ξεκινήσουμε με την αναθεώρηση οδηγίας για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και την υποπτία της αγοράς. Η κυρία Κόμη είναι η συγγετρία και δίνω τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα παρουσιάσω σύντομα την έκθεση που αφορά την ε, γνωμοδότηση για τη γενική ασφάλεια των ε, προϊόντων. Θα σας εξηγήσω λίγο το γενικό πλαίσιο. Η οδηγία για τη γενική ασφάλεια των ε, προϊόντων αφορά την μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας. Πέρσι το 2009 εμείς ε, συντάξαμε μια έκθεση για την εφαρμογή αυτής της οδηγίας, για το τι είχε συμβεί από τον τέχνη. και αναλύσαμε τις βασικές δυσκολίες που υπήρχαν. Όσον αφορά λοιπόν την ε, μεταφορά της στο εθνικό δίκαιο, ε, υπήρχαν κάποιες δυσκολίες, ακριβώς επειδή έχουν κάποιο περιθώριο στη διάθεσή τους τα κράτη-μέλη και βεβαίως ε, υπάρχει και το ζήτημα της εφαρμογής σε σχέση με τα όντως οργανωμένα προϊόντα τα οποία καλύπτονται από την ε, οδηγία. Η κατάσταση λοιπόν δεν ήταν η ίδια σε όλα τα κράτη-μέλη φέτος. Τα πράγματα έχουν αλλάξει και πρέπει να αλλάξει και η οδηγία και ξεκίνησε η Κομισιόν μια διαδικασία διαβούλευσης θα ήθελα να αναφερθώ στα πιο δύσκολα ζητήματα. Τα κριτήρια με βάση τα οποία ένα προϊόν θεωρείται ασφαλές ή όχι. Η χνηλασιμότητα, η λασιμότητα, η από πλευρά κρατών μελών να, ενημερώσουν, να ενημερώνουν την Κομισιόν για τυχόν μέτρα τα οποία περιορίζουν ε, την εμπορία προϊόντων με επικίνδυνες ουσίες. Επίσης, η διαδικασία που θα ορίσει η Κομισιόν για προϊόντα τα οποία περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Επίσης θα ενισχυθεί το σύστημα RAPEX, ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών και θα ε, τυποποιηθεί περισσότερο το σύστημα το οποίο έχουν αναλάβει οι, ευρωπαϊκές, οι ευρωπαϊκοί φορείς τυποποίησης. Έχουμε συζητήσει λοιπόν τα σχετικά. Πέρα από τα γενικά αυτά σχόλια, θεώρησε σημαντικό να καταθέσω και κάποια άλλα ζητήματα για να ενισχύσω το μήνυμά μας. Πρώτα απ' όλα λοιπόν θα ήθελα η Κομισιόν να εξετάσει ένα ενιαίο σύστημα υποπτίας της αγοράς γιατί θεωρούμε πως ε, με την τροποποίηση της οδηγίας και την ε, πιθανότητα εναρμόνισης καλό να έχουμε μία ενιαία φωνή όσον αφορά τη γενική ασφαλή των προϊόντων. Το δεύτερο είναι η χρησιμότητα. Πρέπει οι καταναλωτέ να έχουν τη δυνατότητα να ξέρουν από πού προέρχεται ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, οπότε ζητάμε από την Κομισιόν να κάνει διαβουλεύσεις και αξιολογήσεις αντικτύπου για να αξιολογήσουμε ποια είναι τα κατάλληλα μέσα για να βελτιωθεί η χνηλασιμότητα και ταυτόχρονα να καταπολεμήσουμε το ζήτημα της πειρατείας ε, των προϊόντων. Επίσης υπάρχει το θέμα των ε, μικροτσίπ, ε, ραδιοσυχνοτήτων. Βεβαίω δεν θέλουμε εδώ πέρα να ανησυχήσει κανείς, γιατί έχουμε συζητήσει με τον κύριο Ταγιάννη το κόστος για τις επιχειρήσεις, αλλά ελπίζουμε αυτό να μην έχει αντίκτυπο στους καταναλωτές. και υπάρχει το ζήτημα των νέων τεχνολογιών σήμανσης. Επίσης το σύστημα RAPEX πρέπει να γίνει πιο προσβάσιμο στους καταναλωτές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να είναι ευκολότερο να δουν το τι περιέχεται εκεί πέρα. Και τέλος για το σύστημα τυποποίησης σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να είναι πιο σαφές και να είναι πιο προσιτό για τις ε, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, κυρίως δε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις αυτές όσον αφορά την τυποποίηση και την πιστοποίηση. Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η γενικότερη ασφάλεια των προϊόντων να γίνει πιο εύκολη η διαδικασία πιστοποίησης. Ελπίζω ότι θα συμφωνήσετε με τις γενικές γραμμές ε, της πρότασής μου και βεβαίως είμαι στη διάθεσή σας να ενσωματώσω οποιασδήποτε αλλαγές προτάσεις σας, σχόλιά σας. Γιατί το κύριο μέλημά μας βεβαίως είναι η προστασία των καταναλωτών. Ευχαριστώ. Entschuldigung. Ähm, Entschuldigung, äh, ich wollte fragen, ob es weitere Wortmeldungen gibt von den Kollegen. Ε, με συγχωρείτε. Λοιπόν, ε, υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις από πλευρά συναδέλφων. Κανείς. Α, και αυτό δεν είναι άσχημο. Σας ευχαριστώ πολύ για τη στήριξη. Τότε, επειδή λείπουν οι σχεδόν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 εμπεριστατωμένη δουλειά, συμφωνεί και αυτή με τις δικές μας κατευθύνσεις. Θέλουμε ένα ενοποιημένο σύστημα παρακολούθησης της αγοράς και για μας αλλά και για την σωστή εφαρμογή του. Αλλά δεν... Πρέπει βεβαίως οι κανόνες να περάσουν από τα κοινή μας πίεση στα κράτη-μέλη και στη ΙΜΚΟ. Ο κύριος Χάρμπορ είναι ιδιαίτερος ευαίσθητος σε αυτό. Η χνηλασιμότητα είναι επίσης πολύ σημαντική. Το 2008 με το νέο νομοθετικό πλαίσιο έχει ήδη γίνει πολλή δουλειά γιατί έχουν συμπεριληφθεί νέες διατάξεις συχνηλασιμότητας και με την οδηγία για την γενική οδηγία για τα προϊόντα να ενισχύσουμε το θέμα της συχνηλασιμότητας τώρα όσον αφορά ε, την ιδέα των ISO chips η κυρία Κόμη έθεσε το πιθανό πρόβλημα. Υπάρχει το θέμα του κόστους ε, για τα μικρά ε, αντικείμενα, υπάρχει το πρόβλημα των 50 λεπτών συν ΦΠΑ και υπάρχει το θέμα της εχεμήθειας, της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των δεδομένων. Θα ήθελα να επισημάνω πολύ σωστά, πολύ σύντομα, το θέμα 7 που αφορά τις ποινές. Θα θέλαμε να ήμασταν πιο περιγραφικοί. Εδώ μιλάμε για ναρκοπαίδιο, δεδομένου ότι υπάρχουν εθνικά, νομικά και δικαστικά συστήματα, επί των οποίων δεν έχουμε αρμοδιότητες να επισέλθουμε. Πριν από δύο χρόνια στο πακέτο ε, δεν καταφέραμε πολλά πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε πολύ σαφείς ε, αυτή τη φορά. Κατά τα άλλα, συμφωνούμε με τη συζήτηση που γίνεται σχετικά με την τυποποίηση. Η συζήτηση γίνεται στην Επιτροπή που είναι και η υπεύθυνη Επιτροπή. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εσάς και αν δεν θέλει κάποιος άλλος τον λόγο μπορούμε να τελειώσουμε με αυτό το ζήτημα και να περάσουμε στο σημείο 14. Να υπενθυμίσω πως έχουμε μία μικρή αλλαγή στην προθεσμία για τις τροπολογίες. 16 Νοεμβρίου, 12 το μεσημέρι. Τρίτη, 16 Νοεμβρίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες. Οπότε περνάμε στο σημείο 14, αν συμφωνείτε. Εδώ πέρα μιλάμε για την έκθεση του 2010 αναφορικά με την εφαρμογή των προγραμμάτων της πολιτικής συνοχής. Η κυρία Σούζα Βάγνερ, ο κύριος Σούζα Βάγνερ είναι ο εισηγητής και τον είναι το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. το είπατε και εσείς ο ίδιος ότι πρόκειται για σχέδιο γνωμοδότησης. επί της εκθέσεως ε, της Επιτροπής Ανάπτυξης που είναι αρμόδια επί της ουσίας. Θα σας υπενθυμίσω λίγο το γενικότερο πλαίσιο για ε, τους συναδέλφους που ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Μιλάμε για την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την υλοποίηση των προγραμμάτων 2007-2013 και την πολιτική συνοχή. Αυτή η ανακοίνωση είναι πάρα πολύ σημαντική και σας εξηγώ γιατί. Πρώτη φορά έχουμε μια γενικότερη έποψη εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων συνοχής κατά τη διάρκεια ε, αυτής της φάσης προγραμματισμού, δηλαδή μέχρι το 2013 και βάσει των προγραμματικών ε, εκθέσεων που έχουν εκπονήσει οι χώρες μέλη. Πρόκειται λοιπόν για ένα νέο μέσο το οποίο θα μας επιτρέψει να προσεγγίσουμε την περαιτέρω την πραγματικότητα. Μέχρι τώρα δεν έχουμε ε, βεβαίως πολύ συνολική γνώμη γιατί λίγος χρόνος έχει περάσει αλλά παρόλα αυτά είναι ενδιαφέρουσες ε, οι διαπιστώσεις. Μιλάμε εδώ για πολιτική συνοχή. Ε, πρέπει να ξέρουμε γιατί ακριβώς γίνεται λόγος. Έχουμε εδώ δύο μεγάλες δυσκολίες, δύο μεγάλα εμπόδια στα οποία προσκρούμε. Πρώτον, ο συσχετισμός ανάμεσα στις πλούσιες ε, και τις λιγότερο πλούσιες περιοχές και το δεύτερο εμπόδιο η εξαφάνιση των ανισοτήτων μεταξύ των περιφερειών της Ευρώπης. Για να, ξεπερασ... για να επιτευχθούν οι στόχοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την ολοκλήρωση της Ευρώπης θα πρέπει να ξεπεραστούν τα εμπόδια αυτά. Βεβαίως για να επιτευχθούν οι στόχοι χρειάζεται συντονισμός, χρειάζεται ανταγωνιστικότητα και χρειάζεται και συγκεκριμένο νομοθετικό πλαίσιο. Θα πρέπει λοιπόν να βοηθηθούν οι χώρες μέλη έτσι ώστε να επιτύχουν τους στόχους αυτούς. Ποια είναι τα συμπεράσματα τώρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα οποία αναφέρονται ακριβώς στην ανακοίνωση που ανέφερα εγώ προηγουμένως. Πρώτο συμπέρασμα. πρώτον, θα πρέπει οπωσδήποτε να ε, βελτιωθεί η κατάσταση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα πρέπει η πράσινη πολιτική να μεταφερθεί στην αγορά εργασίας και ε, στην ε, εκπαίδευση καθώς επίσης και στις υποδομές της δημόσιας υγείας. Αυτά είναι σημεία επί των οποίων έχει υπάρξει αρκετή πρόοδος πρέπει να πω αναφέρονται οι πρόοδοι αυτοί και ε, χαιρόμαστε ιδιαίτερος. Δεν μπορούμε όμως να πούμε το ίδιο και για άλλους τομείς. Ακριβώς υπάρχουν κάποια ζητήματα, κάποια σημεία επί των οποίων δεν έχει υπάρξει πρόοδος. Αναφέρομαι ε, σε σημεία όπως η ενέργεια. Στην ανακοίνωση, ας πούμε, λέμε ότι είναι αργή η πρόοδος. 13,2% ε, των ε, πόρων έχουν ε, χρησιμοποιηθεί για την ενέργεια και 20,9% για την αποτελεσματικότητα της ενέργειας. 13 είναι λίγο. Είναι σαφές αυτό. Έχουν υπάρξει βεβαίως ε, πρόοδοι για χώρες οι οποίες ήταν ακόμα πιο πίσω. Και όσον αφορά την ψηφιακή οικονομία, η ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας ε, δεν είναι καθόλου ίδια σε όλες τις ε, χώρες. Για αυτήν έχουν χρησιμοποιηθεί 18,1 των πόρων και για τις τεχνολογίες επικοινωνίας το επίπεδο δεν είναι ομοιογενές και σε γενικές γραμμές παραμένει ακόμα πολύ χαμηλό. Είμαστε εδώ λοιπόν η Επιτροπή Βιομηχανίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ε, κατά την άποψή μας θα πρέπει να εστιαστούμε σε δύο θέματα. Τα εξής. Πρώτα απ' όλα, θα ζητήσουμε από την ε, Επιτροπή οι οικονομίες ενέργειας, οι οικονομίες ενέργειας να εντάσσονται αυτόματα στο τις ε, προϋποθέσεις ε, για τα διαρθρωτικά ταμεία ή τα ταμεία συνοχής. Επίσης, το τμήμα των πόρων που αναφέρονται σε αποταμίευση ενέργειας ή σε χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας θα πρέπει να αυξηθούν. Επίσης, στην έκθεσή μας θα πρέπει να υπογραμμίζουμε την ανισόρροπη ανάπτυξη των επενδύσεων στην ε, ψηφιακή τεχνολογία. Ε, κάτι που αναφέρεται άλλωστε και στην ανακοίνωση τη Επιτροπής και θα ζητήσουμε και από την Επιτροπή και από τα κράτη-μέλη να αυξήσουν ε, την χρηματοδότηση αυτής της τεχνολογίας και της ε, πληροφόρησης και βεβαίως να υπάρξει περισσότερη καινοτομία στον τομέα αυτό, καθώς επίσης και να αυξηθεί ο ρυθμός επενδύσεων στην ευρυζωνικότητα. και θέλουμε η πρόσβαση στο διαδίκτυο να θεωρείται πλέον καθολική ε, ε, χρήση γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καθολική υπηρεσία, συγγνώμη. Σήμερα η πρόσβαση στο διαδίκτυο είναι ένας από τους πιο καινοτόμους στόχους. Η πρόσβαση εννοώ σαν καθολική υπηρεσία. Είναι ένας από τους πιο φιλόδοξους στόχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Μπορούμε να το συγκρίνουμε λίγο με την επανάσταση του υποχρεωτικού σχολείου στην εποχή του Ζιλφερή η μεγάλη καμπή λοιπόν του υποχρεωτικού σχολείου εκείνη την εποχή είναι ε, η δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο για όλους, ε, για τους φτωχούς και τους πλούσιους, για αυτούς που ζουν στην πόλη, στην Ήπεθρο, σε απομακρυσμένες περιοχές, οπουδήποτε και παντού. Εδώ πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας λοιπόν στην έκθεσή μας. Και τελειώνοντας να πω ότι βεβαίως είμαι σε επαφή με τους εισηγητές των άλλων πολιτικών ομάδων και με τους σκιώδεις εισηγητές. Ε, στηρίζομαι ε, στην ε, συνεργασία τους και θα συνεχίσουμε με τη σύνταξη της έκθεσης. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος τον λόγο, τους συναδέλφους. Από ό,τι φαίνεται όχι. Η Κομισιόν θέλει τον λόγο. <coughs> ναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είμαι από την, από την Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον εισηγητή για το σχέδιο προγνωμοδότησης. Είναι ευπρόσδεκτες οι προτάσεις ε, της, του σχεδίου γνωμοδότησης. Μας ικανοποιούν μόνο δύο σύντομες παρατηρήσεις όσον αφορά το θέμα της, ε, των όρων και, ε, και, των, ε, και των προϋποθέσεων. Όσον αφορά την παρούσα ε, προγραμματική περίοδο, οι κανόνες της, των επενδύσεων στην πολιτική συνοχής περιλαμβάνονται στον υφιστάμενο κανονισμό για την πολιτική συνοχής. Ο κανονισμός δεν αναφέρεται στις προϋποθέσεις. Όμως το μελετά το θέμα ε, για το μέλλον η Κομισιόν στις επερχόμενες προγραμματικές περιόδους. Το θέμα ε, αναφέρεται στην έκθεση για τη συνοχή και θα συζητηθεί δημόσια το θέμα τους επόμενους μήνες συμπεριλαμβανομένων και του φόρουμ της συνοχής που θα γίνει το Φεβρουάριο. Άρα η Κομισιόν θέλει να ενισχύσει την ποιοτική απόδοση μέσω την ε, ε, εισαγωγή προϋποθέσεων περιλαμβανομένων και αυτών της ε, εξοικονόμησης ενέργειας. Το δεύτερο ζήτημα που αφορά την αναλογία των επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής, η Κομισιόν αντιμετωπίζει το θέμα σε διμερή βάση με τα κράτη-μέλη. Είναι σημαντικό να πούμε ότι αυτό γίνεται κυρίως ένα κράτος μέλος να πάει στην Κομισιόν και να ξεκινήσει τη συζήτηση αυτή. Άρα είναι θέμα κράτους μέλους. Τα κράτη-μέλη πρέπει να κινηθούν. Μόλις δημιούργησε ένα μέσο η Κομισιόν τεχνικής ε, βοήθειας που θα ε, βοηθά τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν, να υλοποιήσουν τα βασικά τους προγράμματα σε τομείς ε, κλειδιά. Το μέσο αυτό, το εργαλείο αυτό, στόχο έχει τη βελτίωση και της ποιότητας και της ποσότητας του αριθμού των έργων στα πλαίσια αυτά. Αυτές είναι οι δύο παρατηρήσεις μου μόνο σε αυτά που είπατε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ganz herzlichen Dank. Ähm, Wortmeldung sehe ich nicht. Ευχαριστώ, δεν βλέπω κανένα ζητάει το λόγο. Οπότε κάνατε καλή δουλειά. 11 Νοεμβρίου το μεσημέρι είναι η προσημή για τις τροπολογίες, οπότε αν μου επιτρέπετε προτείνω να δούμε το σημείο 15, έτσι ώστε εάν συμφωνεί και ο κύριος Ρέμεκ να συζητήσουμε και αυτό το θέμα τώρα. ε, οι ομάδες να ενημερώσουν και τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Αν ε, λοιπόν δεν υπάρχουν δυσκολίες θα δώσω τον λόγο στον κύριο Ρέμεκ. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Έπληξη μου προκαλεί και είναι και λίγο νωρί ακόμα, αλλά θα δω τι μπορώ να κάνω. Νομίζω πως οι περισσότεροι ξέρετε πως η έκθεσή μου υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό. Οι βοηθή μου και εγώ και άλλοι υποψιαζόμαστε πως η κατάσταση τώρα είναι χειρότερη από ότι ήταν όταν είχαμε ξεκινήσει να ασχολούμαστε με αυτή την έκθεση γιατί τα παλαιά προβλήματα του έργου υπάρχουν, δηλαδή το πώς θα βρούμε τα λεφτά και μετά βέβαια υπάρχει και το ζήτημα του τι θα κάνουμε από εδώ και μπρος με βάση τις ε, πληροφορίες που έχω και έχω πάει σε αρκετές διασκέψεις υψηλού επίπεδου για το θέμα αυτό, έχουν εντύπωση πως κανείς δεν αμφισβητεί το έργο συνολικά. Το έργο είναι κάτι το οποίο ξεκολουθούμε να θέλουμε. Και βεβαίως ε, οι λόγοι για αυτό αναφέρονται στην έκθεση η οποία υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό. Δηλαδή η Κομισιόν θέλει να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητά της έναντι της ε, Ρώσικης Ομοσπονδίας, των ΙΠΑ της Κίνας και άλλων χωρών. Ένα ζήτημα κλείδι κατά την άποψή μου παραμένει το ότι εξακολουθούμε να μην έχουμε βασικές πληροφορίες ε, τις οποίες η Κομισιόν είχε υποσχεθεί εδώ και καιρό. Μέχρι να έχουμε λοιπόν αυτές τις πληροφορίες δεν έχει νόημα να οριστικοποιήσουμε την έκθεσή μας ή και να συνεχίσουμε να ασχολούμαστε με αυτήν. Είναι θέμα της Κομισιόν και στην Κομισιόν βρίσκονται όλες οι ζωτικές πληροφορίες για το έργο αυτό. Ακούσαμε πρόσφατα πως η διαστημική πολιτική θα ενταχθεί σε μια ανακοίνωση για την βιομηχανική πολιτική. Δυστυχώς όμως δεν μπορέσαμε να μιλήσουμε με τον κύριο Επίτροπο, οπότε δεν ξέρουμε. Ένα άλλο κρίσιμο ζήτημα, κατά την άποψή μου, τουλάχιστον έτσι μου φαίνονται τα πράγματα, είναι πως ε, κάποια κράτη-μέλη έχουν νύψει τα σχήρες τους ως προς το έργο αυτό. Αυτό νομίζω είναι αποτέλεσμα και του τι κάνει η Κομισιόν ή μάλλον του τι δεν κάνει και εδώ πέρα μιλάμε για την έλλειψη πληροφοριών. Θα μείνω σε αυτά και ευχαρίστω να απαντήσω σε ερωτήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βεζίνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Πράγματι αναμέναμε τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για το έργο αυτό. Εγώ θα πήγαινα ακόμη παραπέρα και θα ήθελα να ζητήσω μέσω του Προέδρου να γίνει ένα επίσημο ερώτημα προς την Κομισιόν για το τι γίνεται με αυτό το έργο. Εμείς δεν ξέρουμε πού οφείλεται η καθυστέρηση. Μπορεί το πρόβλημα να βρίσκεται στην Κομισιόν, μπορεί να είναι οπουδήποτε. Θα θέλαμε, εν πάση περιπτώσει, να ξέρουμε πού είναι το πρόβλημα. Γιατί αλλιώς δεν θα έχουμε καμία πρόοδο. Σας ευχαριστώ. ο Στουσνόφσκι έχει τον λόγο. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ τίνω να συμφωνήσω με τους ε, συναδέλφους. Όταν ήμουν εισηγητής στο Γαλλιλαίο, η Κομισιόν πάντα έλεγε μέχρι το τέλος του έτους ή αρχές του επομένου έτους θα έπρεπε να είχαμε τις λεπτομέρειες της χρηματοδότησης. Ε, αυτά μας είχε πει η Κομισιόν. Επίσης, μας είχαν πει πως πρέπει να δούμε το ζήτημα της ιδιοκτησίας εδώ πέρα και να δούμε προς τα πού πηγαίνει αυτό το έργο. Έχω την αίσθηση λοιπόν πως ε, με τα νέα διοικητικά του Γαλιλαίου έχουμε μια στασιμότητα γιατί δεν υπάρχει απαραίτητη στήριξη από την Κομισιόν. Στηρίζω λοιπόν αυτό το οποίο ζήτησε ο κύριος Ρένοκ, πράγματι να υπάρχει μια καλή έκθεση αλλά και να ξέρουμε πού πάνε αυτά τα έργα και ποιο θα είναι το αποτέλεσμα πέρα από το 2013 και 2014 χρειαζόμαστε αυτές τις λεπτομερείς πληροφορίες. Και ξέρετε πως ε, αυτά τα, 2000, ε, αυτά τα στοιχεία του 2012 είναι πάρα πολύ σημαντικά πριν ξεκινήσει να λειτουργεί το σύστημα. Ή λοιπόν που δεν ήρθε ο κύριος Επίτροπος σήμερα, γιατί ο κύριος Επίτροπος θα μας έδινε σημαντικές πληροφορίες. Ακούσαμε και στο παρελθόν στην Επιτροπή μας πώς θα μας έδιναν τις διοικητικές και οικονομικές πληροφορίες. Πρέπει να τα έχουμε αυτά, αλλιώς δεν ξέρουμε πού πηγαίνει αυτό το έργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάποιος άλλος θέλει τον λόγο. Είναι κάποιος εδώ από την Κομισιόν. Θέλετε τον λόγο. Παρακαλώ. Με μικρόφωνο παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, εκπροσωπώ το Γενικό Γραμματέα. Ε, εάν ε, είχε τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα στις 11 η ώρα, νομίζω θα ήταν ε, εδώ πέρα ένας ειδικός σας απαντήσει. Δυστυχώς όμως δεν είναι εδώ. Σημειώνω τα σχόλιά σας και θα επανέλθω αργότερα. Ευχαριστώ. Ωραία, σας ευχαριστώ. Κύριε Ρέμεκ, θέλετε πάλι τον λόγο. Ευχαριστώ. Ε, δεν είναι η πρώτη φορά που στην περίπτωση ενός έργου ορόσημου της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδιαφέρει ολόκληρο τον κόσμο, εμείς πηγαίνουμε ε, Δεν μας ωφέλει αυτό. Έχω δει και ξαναδεί την κοινή γνώμη στην Ευρωπαϊκή Ένωση να στρέφεται κατά αυτού του έργου, γιατί κανείς δεν ξέρει τίποτα και δεν μπορεί να μάθει τίποτα γι' αυτό. Υπάρχουν διάφορε διάφορες διαρροές, σκεμμένες ή που υπονομεύουν το έργο και είναι κρίμα γιατί είναι παραπλανητικά όλα αυτά. Στην καλύτερη των περιπτώσεων είναι κρίμα το ότι δεν έχουμε καταφέρει να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα με έναν τρόπο ε, πιο ήρεμο και σε ένα περιβάλλον πιο ήρεμο. Δεν ξέρω, ίσως να μην έχει κανείς άλλος να πει τίποτα από ε, αυτού, αλλά θα μου προξενούσε εντύπωση. Οπωσδήποτε ευχαριστώ τους συναδέλφους που έλαβαν το λόγο για να με στηρίξουν. Και νομίζω πως θα συμφωνήσω το πάρει με τον κύριο Μπρεζίνα. Είναι καλή ιδέα να βρεθούμε με τους σκιώδεις συζητητές και να προτείνουμε μια λύση στους συναδέλφους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. αντιλαμβάνομαι αυτά τα οποία είπατε. Πραγματικά δεν είναι δυνατόν. Νομίζω κύριε Ρέμεκ την πρόταση του κυρίου Βρεζίνα πρέπει να την ε, υιοθετήσετε, να συναντηθείτε οι συγητές και οι και να κάνω και εγώ μια πρόταση. Εάν συνεννοηθείτε, ε, μπορείτε να, να γράψετε μια επιστολή, να απευθύνετε μια επιστολή στον κύριο Ταγιάννη και μπορώ και εγώ να σας υποστηρίξω. Αρκεί να συμφωνείτε, γιατί εδώ και μήνες πάει μπρο πίσω αυτή η υπόθεση, δεν υπάρχει καμία πρόοδο. ε, πρέπει να στείλουμε ένα μήνυμα. Πρόταση λοιπόν. Σκεφτείτε το μαζί, εγώ είμαι διατεθειμένο, είτε μόνο μου ή όλοι μαζί, να απευθύνουμε μια επιστολή για να ασκήσουμε την απαραίτητη πίεση. Συμφωνείτε? Ωραία. Σας ευχαριστώ λοιπόν. Θα παρακαλέσω την ε, γραμματεία να κινήσει τη διαδικασία. Οπότε τελειώσαμε και με το σημείο 15 και έχουμε λίγη ώρα γιατί η ψηφοφορία είναι στις 10. Οπότε μπορούμε να πάμε όλοι για ένα καφεδάκι, αλλά σας παρακαλώ 10 η ώρα στην ώρα μας εδώ πέρα για να ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ.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 Meine, Συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι, περνάμε στις ε, ψηφοφορίες, οι οποίες είναι και σημαντικές και πολύπλοκες σήμερα, οπότε θα ήθελα να με ακούσετε λίγο, δύο-τρία λεπτά, γιατί υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να ανακοινώσω. Πρώτα απ' όλα, μετά τις ε, ψηφοφορίες θα ξαναπεράσουμε στο σημείο 15 για το διάστημα, γιατί μεταξύ ήρθε εκπρόσωπος της Κομισιόν και θέλω να δώσω στην Κομισιόν την ευκαιρία να μας πει κάποια πράγματα για αυτό το ζήτημα, γιατί είχαμε μια ευρύτατη συζήτηση με ερωτήματα τα οποία έμειναν ανοιχτά. Μετά τις ψηφοφορίες λοιπόν θα ήθελα να παρακαλέσω όσοι άλλοι θέλουν να βγουν έξω να φύγουν γρήγορα και όσοι ενδιαφέρονται για το θέμα να μείνουν για να μπορέσουμε να συζητήσουμε με την Κομισιόν για το θέμα αυτό. Δεύτερη παρατήρηση. Και ζητώ την προσοχή σας λίγο. Χθες 8 ή 9 η ώρα το βράδυ έλαβα τους καταλόγους της ε, ψηφοφορίας και 9 ή 10 τον κατάλογο της ομάδας μου, της κάθε ομάδας. Δεν θέλω να πω γιατί είναι έτσι τα πράγματα και πώς είναι έτσι. Ένα πράγμα μόνο. Στην επόμενη ψηφοφορία, ό,τι έρθει αργά το βράδυ δεν θα τεθεί σε ψηφοφορία. Θα αναβληθεί η ψηφοφορία και θα σας πω γιατί. Για εμένα ήταν δύσκολο ως πρόεδρος που είχα τη βοήθεια να τα δω όλα αυτά. Οπότε είμαι σίγουρος για έναν απλό συνάδελφο που έχει έρθει σήμερα να ψηφίσει πως είναι αδύνατον αν έρχεται το βράδυ ο κατάλογος της ψηφοφορίας να μπορέσει να ψηφίσει το άλλο πρωί σωστά. Είναι αδύνατον και δεν θέλω να αναγκάσω κανέναν άνθρωπο, ούτε να κατηγορήσω κανέναν, ούτε βουλευτή, ούτε συνεργάτη. Αλλά θα πρέπει πραγματικά να μπορέσουμε να, να δούμε και αυτούς τους καταλόγους των ψηφοφοριών. Οπότε θα πρέπει να είναι στη διάστηση των συναδέλφων από το απόγευμα της προηγουμένης. Εάν δεν γίνει αυτό θα αναβληθεί η ψηφοφορία. Έτσι θα γίνει, δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Ήμουν έτοιμος να το κάνω και σήμερα αυτό, αλλά είναι σημαντικά αυτά τα θέματα και βιαζόμαστε. Και είναι και ιδιαίτερη αυτή η εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα έλειπαν οι συνάδελφοι. Ζητώ λοιπόν λίγη κατανόηση. Ε, δεν είναι καλό να φερόμαστε έτσι ο ένας τον άλλον. Αυτή είναι η δεύτερη παρατήρηση που ήθελα να κάνω. Η τρίτη παρατήρηση. Θέλω λίγο την κατανόησή σας. Έχουμε πάλι ένα κατάλογο με πολλές και πολύπλοκες ψηφοφορίες. Έχουμε το πρόβλημα σήμερα πως πρέπει να μάθουμε και το πώ λειτουργούν τα μηχανήματα. Ο Λούις ο μόνος από τη γραμματεία που ξέρει πώς να χειρίζεται αυτή τη συσκευή λείπει. Εγώ πλέον δεν το καταλαβαίνω, αλλά δεν χρειάζεται για να το καταλάβω. Προσπαθήσαμε λοιπόν να το οργανώσουμε. Παρακαλώ, έτσι, λίγη υπομονή σήμερα παραπάνω. Και ο κύριος Τούμες ζήτησε τον λόγο επί της διαδικασίας. Παρακαλώ λοιπόν. Ε, πρόεδρε, δεν νομίζω ότι είναι σωστό να παίρνουμε τόσο αργά τους καταλόγους ψηφοφοριών και να τεθεί το θέμα στην επόμενη συνεδρίαση των ε, συντονιστών, να έχουμε αναλύσεις. Και όταν υπάρχουν εκθέσεις για τις οποίες γίνονται ε, τεχνικές συνεδριάσεις στο προσω... στα... ανάμεσα στα μέλη του προσωπικού, να μας τα στέλνουν γέρος. Για άλλες για άλλες ψηφοφορίες και για λόγους που δεν θέλω να επισέλθω εδώ, όταν δεν γίνεται σε άλλες πολιτικές ομάδες συνεδρίαση ε, του προσωπικού. Δίνονται ελάχιστο, δίνεται ελάχιστος χρόνος στους εισηγητές και τελικά υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση και πολύ στρες στο τέλος. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το συζητήσουμε με τους συντονιστές γιατί πρέπει να λυθεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και για τη στήριξη. Ο κύριος Οντή. Κύριε Πρόεδρε, συμφωνώ με αυτά που ακούστηκαν και να πω επίσης ότι το σύνολο διαπιστώνομαι υποβάθμιση της κοινοβουλευτικής εργασίας. Κάποια στιγμή θα μας κατηγορήσουν οι πολίτες μας ότι ψηφίζουμε οτιδήποτε χωρίς να το καταλαβαίνουμε. Και όσον αφορά τα συμβιβαστικά κείμενα, πολύ αργά έφτασαν, φτάνουν στα κείμενα αυτά και ε, λανθάνουν οι συντονιστές όταν δέχονται αυτές τις συμβιβαστικές Όσον αφορά την πολυγνωσία έχουμε πρόβλημα ε, και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε λίγο πιο σοβαρά την κοινοβουλευτική μας εργασία. Ευχαριστώ πολύ και να είστε σίγουρος πως θα το συζητήσουμε. Έτσι θα γίνει την επόμενη φορά όπως σας είπα. Λοιπόν, ας προσπαθήσουμε τώρα να περάσουμε στα συγκεκριμένα θέματα. Πρώτη ψηφοφορία αφορά το, τα ανθρακοριχεία, την έκθεση Ζαντό. Τα έγγραφα τα έχετε και τον κατάλογο. Ξεκινάμε λοιπόν. Οπότε, ψηφίζουμε την τροπολογία 28 υπέρ. Κατά. Εποχές γκρίνεται. 66 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 69 υπέρ. Εάν απορριφθεί. Όχι, την ψηφίζουμε κανονικά. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 70 υπέρ. Κατά. Να το ξαναδούμε. 70 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 71 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται 72 όχι κατά καταπίπτει 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 1 υπέρ κατά εποχές εγκρίνεται. Να επαληθεύσουμε. Συμβαστική 1. Ναι. Να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία πρώτα, λόγω του τεχνικού προβλήματος. Όχι, δοκιμαστική. αν είναι ωραίος ο καιρός, ναι ή όχι. Είναι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Τώρα είναι εντάξει. Και τώρα ψηφίζουμε τη συμβαστική 1, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. και το αποτέλεσμα είναι σαφές. Δεκτή λοιπόν. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 86, α ήταν ταυτόσημη. 84 υπέρ. Με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. 84 με την προφορική τροπολογία υπέρ. Κατά. Ε, δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Η 84 με την προφορική τροπολογία. Με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Είναι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Εγκρίνεται λοιπόν. 83 με την προφορική τροπολογία. Καταπίπτει. 16 λοιπόν υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 87 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 88 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 3 υπέρ. Κύριε Μακινκέβιτς, υπάρχει κάποιο πρόβλημα? Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θέλω να φύγει η λέξη only από τη συμβιβαστική πρόταση. Στη δεύτερη παράγραφο. Στην συμβιβαστική τρία. Υποθέτω πως έχετε συμφωνήσει συμφωνείτε με αυτό το οποίο λέει ο συγητής εδώ πέρα να φύγει προφορική τροπολογία η λέξη only. Λοιπόν, με ναι, αυτή τη μικρή αλλαγή, η συμβαστική τρία, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 85 υπέρ. 85 υπέρ. Α, συγγνώμη. Συγγνώμη, συγγνώμη, 95. Δικό μου λάθος. Νούμερο 95 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 100 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε την 100 Άρχιε τη ψηφοφορία πέρασε και εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Εκατόν ένα. Εκατόν ένα υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 20 καταπίπτει. 103 υπέρ. Κατά αποχέση. Εγκρίνεται. 104 καταπίπτει. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 105 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ναι, να υπαλληθεύσουμε, να υπαλληθεύσουμε. 24. Και πέρας. Δεκτή. 107. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 25 υπέρ κατά αποχές δεν, δεν βλέπω, με συγχωρείτε, πρέπει να την επαναλάβουμε 25 υπέρ 25 25 παρακαλώ, όσοι είναι υπέρ, κατά. Αποχές. Ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία, συγγνώμη. 25 υπέρ. Να έρχεται η ψηφοφορία, μάλλον. Πέρας. Δεκτή. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 108 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 109 υπέρ καταπίπτει συγγνώμη και 110 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 111 13 14 υπέρ κατά αποχές θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά δεν μπορώ να διακρίνω. Άρχη η ψηφοφορία. 112, 13, 14. Πέρας. ενα παραπάνω από το ΕΛΚ. Ε, να την επαναλάβουμε. Συγγνώμη. Έγινε ένα λάθος. Πρέπει να επαναληφθεί η ψηφοφορία. 112, 13, 14. Άρχεται η ψηφοφορία. Λοιπόν, εγκρίνεται. Περνάμε στην 29 υπέρ. Κατά. Ξανά. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 30 υπέρ. κατά αποχές επαλήθευση ε, συγγνώμη δεν, δεν μπορώ να διακρίνω 30 λοιπόν να έρχεται η ψηφοφορία Όλα εντάξει. Απορρίπτεται. 30 λοιπόν υπέρ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη. 31 και 32 καταπίπτουν, 2 καταπίπτει. 31 muss abgestimmt werden, weil 30 abgelehnt worden ist. Dankeschön. Ich Πρέπει να ψηφιστεί 31. Λοιπόν, συγγνώμη, κάνω λάθος. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. Την 31 ψηφίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Πέρας εγκρίνεται. 32 Πρέπει και αυτή να ψηφιστεί. Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Κανείς από τους Σοσιαλδημοκράτε. 32 ξανά. 32 ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση. Συμβαστική 5 άρχιτη ψηφοφορία. Δύο παραπάνω από το ΕΛΚ. Ξανά λοιπόν. Τώρα Ξαναψηφίζουμε. Υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα. Άρχιε τη ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 27 υπέρ, 25 κατά, μία αποχή. Περνάμε στο 33. Τροπολογία 33. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 34. Όχι. Ναι. 34. Α, και οι 35 καταπίπτουν. Περνάμε στην υπαριθμόν 3 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. 36 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. Συγγνώμη. 36. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Εντάξει. 27 με 27 απορρίπτεται. Συμβιβαστική 6. Υπέρ. Κατά. Εποχές Απορρίπτεται. Ε, ήταν σαφές. Ε, ήταν σαφές νομίζω. Θέλετε να παληθεύσουμε. Ωραία. Παληθεύσουμε την συμβαστική 6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ε, σαφές. 37. Υπέρ. Κατά. Αμποχές. Απορρίπτεται. 41. Μια στιγμή. 41 και 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 39 υπέρ. Α, καταπίπτει. Καταπίπτει. Είναι πολύπλοκα γιατί δεν, είναι, δεν αφορά μόνο τις συμβαστικές τροπολογίες αλλά την κάθε τροπολογία. Λοιπόν, 40 πίπτη. Περνάμε στην 4 λοιπόν. Και αυτή. 42. Τη 42 θα ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Σα ε, σας παρακαλώ να σηκώνετε τα χέρια σας. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε συμβαστική 7. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται με ισοψηφία. Οπότε περνάμε στην 45 υπέρ. Κατά. Ξανά. 45 υπέρ. από δεν ψηφίζουν. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 48 και 49 ταυτόσημες. Υπέρ. Κατά εγκρίνονται 50 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε 53 υπέρ άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 52 ως προσθήκη. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική 8. Υπέρ. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Γκρίνεται. Άμα I think number Exactly. Νομίζω ότι περνάμε στην 9. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 64 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 11 υπέρ να, να επαληθεύσουμε να, να την 64 άρχεται ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται ευχαριστώ 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 65 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 υπέρ. κατά καταπίπτει. Οπότε περνάμε στην τελική ψηφοφορία για... Α, ο κύριος Ζοντό. Ναι, παρακαλώ. Euh, euh, Κύριε Πρόεδρε, η εξαιρετικά κοινωνική, πολιτική, ε, πολιτιστική και οικονομική διάσταση είναι δεδομένη, αλλά όσον αφορά η αύξηση των δαπανών ε, είναι ανεύθυνη όχι μόνο από δημοσιονομική άποψη αλλά από ε, περιβαλλοντική και οικονομική άποψη και γι' αυτό δεν θα ήθελα το όνομά μου να συνδεθεί με αυτό. Ευχαριστώ. Ωραία. Το λαμβάνουμε υπόψη. Ψηφίζουμε λοιπόν το σύνολο της έκθεση με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία και πέρασε. Ωραία, εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Έγινε δεκτή. βέβαια ποιον συγχαίρω. Εν πάση περιπτώσει. Περνάμε στο σημείο 8. Ενεργειακή αποδοτικότητα. Την έκθεση την έχετε. Τώρα είναι ακόμη πιο πολύπλοκη. Οπότε θέλω και εδώ τη βοήθειά σας. Ξεκινάμε. Όχι. 63 πρώτα απ' όλα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 83 υπέρ. Πέφτουν, καταπίπτουν οι υπόλοιπε. Λοιπόν, 83. Ε, να ψήσουμε ηλεκτρονικά. Κατευθείαν, κατευθείαν. Άρχεται τη ψηφοφορία. Γιατί θα είναι και τσίμα τσίμα. Και πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 8 υπέρ Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 8 συν 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 89 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε το 89 έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απορρίπτεται. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 107 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 114. Χωριστή ψηφοφορία. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές. Δεν έχω ιδέα. Λοιπόν, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Το δεύτερο μέρος 114 αρκετή ψηφοφορία. Και πέρας είναι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. 27 με 27 απορρίπτεται. 12 συν 1 υπέρ. Α, συγγνώμη. 116 πρώτα. 116 υπέρ. Κατά. Αποχές συγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 συν 1 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 90 καταπίπτει 90 Θέλετε την, την 12 συν 1 να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία και πέρας όχι απορρίπτεται απορρίπτεται σαφές οπότε πάει και η 90. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 91 ψηφίζουμε χωριστά. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτονται Συμβαστική 15 υπέρ. Να επαληθεύσουμε τι... την 91. 91 λοιπόν άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρασε. Απορρίπτεται. Συμβαστική 15. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει. 122 πρέπει να την ψηφίσουμε. Λοιπόν, σε δύο μέρη. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο τμήμα Λοιπόν, επαλήθευση. 122 πρώτο μέρος. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. Απορρίπτεται. Ορίστε. 26 έναντι 26 και 0 αποχές. Απορρίπτεται. Περνάμε στο δεύτερο μέρος. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 123 καταπίπτει. 124 ψηφίζεται. Λοιπόν, 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 συμβιβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 17 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 150 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 157 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ, Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 168 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 182 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 186 πέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να επαληθεύσουμε 186. Άρχεται η ψηφοφορία. Και πέρας. Δεκτή. Η 186. Περνάμε στην 187 υπέρ. Κατά. Ε, ε, συνάδελφοι, φωνάζετε επαλήθευση. δεν έχω πει τίποτα και φωνάζετε... Ε, δεν είναι δυνατόν. Λοιπόν, σηκώστε τα χέρια ψηλά να γίνουν πιο εύκολα τα πράγματα. 187, ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Τώρα νομίζω είναι δεκτή. Τώρα να επαληθεύσετε, εντάξει, το καταλαβαίνω. Λοιπόν, 187. Άρχεται. Και πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 21 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 194. Καταπίπτει. Συμβαστική 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 211 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 26 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 225 υπέρ κατά αποχές δεκτή καταπίπτει επόμενη συμβαστική 27 υπέρ κατά αποχές δεκτή 233 υπέρ κατά αποχές δεκτή 234 σε τρία μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές. Να επαληθεύσουμε το δεύτερο μέρος, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Τρίτο μέρος, υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 98 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές Τι Δεύτερο μέρος. Καταπίπτει. 238. Θέλει να πει κάτι ο εισηγητής. Για τις ε, παραγράφου, για τις ε, τροπολογίες 238 ε, αναφέρεται ότι καλύπτονται από τον συμβιβασμό του 28. Οπότε τέλος δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε άλλο με αυτό και περνάμε κατευθείαν στην Συμβιβαστική 29. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 282 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 253 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Περνάμε 254, 55, 56 και 57. Ποιο είναι υπέρ ταυτό μα. Κατά. Αποχέ. Δεκτή. Συμβαστική 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 31 συν 1. Πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, 31 συν 1. Ποιο είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 272 ως προσθήκη. Κύριε Μπέντσεν. Και εδώ, επί της διαδικασίας καλύπτεται από την τροπολογία 32. Ευχαριστούμε. Οπότε δεν ασχολούμαστε και με αυτό. Ο κύριος Ζαντό διαφωνεί, οπότε έχει το λόγο. Λυπάμαι κύριε Πρόεδρε. Αμφισβητώ. Δεν νομίζω ότι καλύπτεται η τροπολογία. Καλώς. Τι θα γίνει τώρα. Ο ένας λέει πως καλύπτεται, ο άλλος όχι. Είχαμε και την προηγούμενη φορά το ίδιο θέμα τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση. Πρέπει να ξεκαθαρίσει. Ε, εγώ, θεωρώ πως πρέπει να ψηφίσουμε. Αν επιμένει αυτός ο οποίος κατέθεσε την τροπολογία, νομίζω πως πρέπει να την ψηφίσουμε, αν συμφωνείτε. Λοιπόν, 272, τι ψηφοφορία. Σε ψηφοφορία. 272. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Και λύθηκε το πρόβλημα. 284 καταπίπτη. Όχι. 284, 85 και 86 μπορούμε να τις δούμε μαζί. Να τις ψηφίσουμε όλες μαζί. Ναι. 84, 85 και 86 ως προσθήκη. ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Οπότε απορρίπτονται. Συμβαστική. Α, να επαληθεύσουμε. Συγγνώμη. 84, 85, 86 ως προσθήκη. Άρχεται τη ψηφοφορία. Πέρας. Α, Δεκτέ. Ε, μία ψήφο διαφορά. Ωραία, σα ευχαριστώ. Συμβαστική 32 είναι 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 33. Υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 34 υπέρ. Κατά αποχές Συμβαστική 35, όχι. Ναι, 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 301 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε. 301. Άρχεται η ψηφοφορία. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Πέρας. Δεκτή. Οπότε περνάμε στην συμβαστική 36. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 37. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. το δεύτερο τμήμα της 311. Θα το ψηφίσουμε. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Προφορική τροπολογία. Θα επαληθεύσουμε το δεύτερο τμήμα της 311 με την προφορική τροπολογία. Α, όχι. Όχι, όχι, χωρίς. Μόνο το δεύτερο τμήμα της 3.11. Άρχεται η ψηφοφορία. And closed. Και πέρασε. Και γίνεται δεκτή. Περνάμε στην πρόταση του εισηγητή για προφορική τροπολογία. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Δεκτή. Όχι, 312. 312 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. 312. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Ε, συγγνώμη, αλλά καμιά φορά δεν μπορώ να καταλάβω ότι ψηφίζεται. Συμβαστική 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 321 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. 321. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 322 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 324 υπέρ. Κατά. Να, πήγα πολύ γρήγορα. 324 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 325 υπέρ κατά αποχές δεκτή 39 συμβαστική υπέρ κατά αποχές δεκτή 328 υπέρ κατά επαληθεύση 328 άρχεται η ψηφοφορία Απορρίπτεται. 3.29 πρέπει να ψηφιστεί υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 329. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε όλοι παρακαλώ. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 41 υπέρ. Κατά. Αποχές Συμβαστική 40 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτεί. 334 αποσύρθηκε. 337 υπέρ. 337, 337 υπέρ. Κατά. Αποσύρθηκε η 334. Λοιπόν, η 337 γίνεται δεκτή. Συμβιβαστική 42 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 339 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 343 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 344 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος καλύπτε. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 346 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Συμβιβαστική 43 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 349 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 45 υπέρ κατά αποχές συμβιβαστική 46. Παρακαλώ, κύριε Μπέντσον. Ε. Για την 364, παράγραφος 35α, καλύπτεται από το συμβιβασμό 39. Okay. Ωραία. Άρα περνάμε στη συμβαστική 46. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 371 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 372 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. 372. Άρχεται η ψηφοφορία και πέρασε. Και απορρίπτεται. 373 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ναι. Ποιος είναι υπέρ. 373. Κανείς. Ευχαριστώ. Κατά. Αποχές δεκτή. 375. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Να την παληθεύσουμε. Τα ωραία. 3,75 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Και έγκαιτα. Ε, καμιά φορά είναι μία ψήφωση διαφορά. Καλό είναι να σηκώνετε τα χέρια σας ψηλά. 376 υπέρ 376 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 378 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 379 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 385 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος πέρ. δύο μεγάλες ομάδες ήταν. Λοιπόν, να επαληθεύσουμε το πρώτο μέρος της 385. Άρχεται η ψηφοφορία και πέρασε. Απορρίπτεται. Δεύτερο μέρος πέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 47 υπέρ, κατά αποχές Συμβαστική 48 υπέρ, κατά αποχές Τι; 3.97 υπέρ, κατά αποχές. Να επαληθεύσουμε. 3.97. Άρχεται η Πέρασε. Έχει λήξει η ψηφοφορία. Η Δερμηνία ακούγεται, δεν μπορεί να παρακολουθήσει τον πρόεδρο. Λοιπόν, επαναλαμβάνω την ψηφοφορία γιατί πήγα πολύ γρήγορα και κάποιοι ψήφισαν λάθος. 397. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονική. Πέρασε. Απορρίπτεται. Α, άξιζε τον κόπο. Λοιπόν, περνάμε στην 402. Όχι 400. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 402 καταπίπτει, οπότε περνάμε στη συμβαστική 49. 49 βλέπω εγώ. Λοιπόν, ποιος είναι υπέρ τη συμβαστικής 49. Κατά. Αποχές. Κτή. 410 υπέρ. Κατά. Α, πολύ γρήγορα. 410 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 4-11 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 4-12 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 413 υπέρ. Κατά αποχές. Απορρίφτεται. 414 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 415 υπέρ. 414. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 415 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 416 υπέρ. Όχι, δεν είναι δεκτή 414, οπότε 416 υπέρ. Κατά. Δεν ψηφίσετε. 416. Ποιος είναι υπέρ, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κατά. Ε, πάλι δεν βγάζει συμπέρασμα. Λοιπόν, να επαληθεύσουμε. Να αρχίσει η ψηφοφορία. Ένα παραπάνω από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ. Και απορρίπτεται. 4-17 υπέρ. Κατά. αποχες ακτη Δεκτή. 4-18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μπορούμε να την παλήθευσουμε λοιπόν την παλήθευση 4-18 Πέρας. Δεκτή. 4-20 υπέρ. Ναι, γιατί έφερε κάποιον μέσα ο κυριος Τούρμες. Λοιπόν, 4-20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Νομίζω ήταν σαφές. Λοιπόν, 4-20 επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτή. Έχετε δίκιο. Λοιπόν, 4-24 πέρα. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 1. Ε, πρέπει να παραγγείλουμε μεσημεριανό μου φαίνεται. Συμβαστική 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ε, απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική Λοιπόν, 16. Να την επαληθεύσουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές Προφορική τροπολογία στην 20 υπέρ. Ναι, ένα λεπτάκι. Ο κύριος Βιντάλ το λόγο. Όταν ψηφίζουν όλα τα μέλη, τα παρόντα μέλη, ε, και ξέρουμε ότι έχουν δικαίωμα, <clears throat> ποιος ε, ε, είναι ο αριθμός του συνόλου των, ψηφισμά, των ψηφισάντων ποιοι έχουν ε, δικαίωμα ψήφου. Δηλαδή, ε, από όλε τι πολιτικέ ομάδε, ποιο είναι ο αριθμό των ψηφισάντων που πρέπει να βλέπουμε στι οθόνε μα. Κανονικά 53, αλλά κυμαίνεται. Δεν ψηφίζουν όλοι οι συνάδελφοι. Ε, δεν μπορώ να το αλλάξω εγώ. Καμιά φορά δεν ψηφίζουν όλοι οι συνάδελφοι. Σήμερα ήταν 53. Όταν ψηφίζουν όλοι, 60 είμαστε λέει ο πρόεδρος κανονικά. Όχι. Α, εδώ μου δίνουν τις πληροφορίες. 55. 55 είναι ο κανονικός αριθμός, αν είναι όλοι παρόντες. Τα τελευταία λεπτά το υψηλότερο που επιτύχαμε ήταν 53. Οπότε 2 δεν είναι εδώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο κύριος Βεθαλκόδρας. Λοιπόν, συμβαστική 1. Ξαναψηφίζουμε. Υπέρ. Α, συγγνώμη. Έχω αρχίσει και μπερδεύομαι. Ναι. συγχωρείτε. Λοιπόν, ήμασταν ναι, στην 20 με την προφορική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συνδεστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Να την επαληθεύσουμε. Πάντα στι δικέ μου θέλετε επαληθεύσει. Λοιπόν, 24, να την επαληθεύσουμε, είπε, ε, η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι οι συνάδελφοι. Πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 36 σε δύο μέρη. Πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτή. Δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 37, 38, 39 υπέρ Κατά. Να επαληθεύσουμε. 37, 38, 39. έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Δεκτές. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική έξι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. 44 ε, υπέρ. Ε, όχι. 44 άρχεται η ψηφοφορία. Closed. Πέρας. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Να επαληθεύσουμε. η ψηφοφορία επί της 45. Πέρας. Δεκτή. 46 καταπίπτει, 47 υπέρ. Κατά. Και οι υπόλοιποι. Ε, απεργία. Λοιπόν, δεκτή. Συμβαστική έξι είναι ένα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 48 μέρος πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. Δεύτερο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω απορρίπτεται. Ποιος φωνάζει να επαληθεύσουμε. να επαληθεύσουμε. Το δεύτερο μέρος άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 55 καταπίπτει, 56 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 57 προφορική τροπολογία, τι είναι αυτό, 57 προφορική τροπολογία υπέρ. Πάλι ρεμπιχ, έχεις τον λόγο. Είναι η τροπολογία μου και νομίζω ε, είναι πάρα πολύ αυστηρό εδώ πέρα, το ΣΑΜ, οπότε είμαι κατά της προφορικής τροπολογίας. Οπότε ψηφίζουμε την αρχική ε, διατύπωση, ποιος είναι υπέρ, χωρίς την προφορική τροπολογία. Υπέρ, κατά αποχές, δεκτή. Όχι. Λοιπόν, η 57 του συναδέλφου Ρούπη χωρίς την προφορική τροπολογία άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Με ισχυρή μειοψηφία. 58 πάει, 59 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 60 καταπίπτει. Όχι, 60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Να παληθεύσουμε την 60, άρχεται η ψηφοφορία. Δεχθεί. Απορρίπτεται με ισοψηφία. 61 πίπτη. ψηφίζουμε την 62 υπέρ. Κατά αποχές δεχθεί. Παριθμόν 1. Όχι, δεν χρειάζεται να το ψηφίσουμε. 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 2 καταπίπτει. Τώρα 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Όλες μαζί υπέρ κατά αποχές δεκτή. Ένα του περιβάλλοντος καταπίπτει, δύο το ίδιο, τρία το ίδιο, τέσσερα, Ψηφίζουμε την 4 του περιβάλλοντος. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Κατά. αποχέ, Απορρίπτεται. 5 NV καταπίπτει. Ε, 6 ε, ναι. του περιβάλλοντος υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 7 περιβάλλοντος υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 NB υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 του περιβάλλοντος υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 περιβάλλοντος υπέρ κατά αποχές δεκτή Δεκαοχτώ, όχι καταπίπτει. 19 δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτή 22 καταπίπτη 23 υπέρ κατά σας παρακαλώ λοιπόν 23 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε. 23. Πέρας. Δεκτή. 24 υπέρ. Κατά. Εποχές. Απορρίπτεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 30 υπέρ κατά αποχές 30 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή 35 υπέρ κατά αποχές δεκτή περιφερειακή 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή και περνάμε στην τελική ψηφοφορία, άρχιτη ψηφοφορία. Και πέρασε. Ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Ξαφνικά έχουμε 54 εδώ Λοιπόν, δεκτή με μεγάλη πλειοψηφία συγχαρητήρια. Περνάμε στην επόμενη έκθεση. Έκθεση δηλαδή για το ΑΕΠ της κυρίας Ματίας. Περνάμε συμβαστική 1 υπέρ. Τρία Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 26 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 33 υπέρ κατά αποχές δεκτή 34 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 6 υπέρ ε μα κακία το κάνετε με τις δικές μου λοιπόν 34 παλήθευση 34. τέσσερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. M. Έχουμε πραγματικούς φίλους στην αίθουσα. Λοιπόν, συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 38 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, δεκτή, συγγνώμη. 39 υπέρ κατά έχεις δεκτή 40 υπέρ κατά αποχές δεκτή απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή 53 υπέρ κατά αποχές Λάθος. Μπερδεύτηκα λίγο. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 Μάρκος Πίπερ συγγνώμη για τον κατάλογο συμφωνίων του ΕΛΚ να πω ο κύριος Τσουκαλάς ο ε, μου εξέθεσε περαιτέρω επιχειρήματα θέλω να συστήσω στο ΕΛΚ να υπερψηφίσει την υπαριθμόν 20, καθώς στον κατάλογό μας είναι ένα μείον. Ωραία, περνάμε στην 20, Ποιο είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή τελική ψηφοφορία άρχεται πέρασε Αποχές. Ευχαριστώ. Συγχαρητήρια. Περνάμε στην εκθεσή Τικάου. Μαύρη θάλασσα. Συμβαστική 1 υπέρ. Κατά. Αποχές δεχτεί. 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεχτεί. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεχτεί. 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική 5. Υπέρ, πάτε κατά αποχές δεκτή. 15. Καταπίπτει. Αχα. 20 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 21 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ. Κατά αποχές. Να επαληθεύσουμε. 22. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Δεκτή. 23 πέρα Κατά. Αποχές. Δεκτή. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 26 υπέρ, κατά αποχές 27 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 28 8 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 29 υπέρ, κατά αποχές 30 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 31 καταπίπτει, 32 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 33 υπέρ. Κατά. Κατά. χέρι δεκτεί? 34 υπέρ. Κατά. χέρι. Απορρίπτεται. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 36 υπέρ. Κατά. χέρι δεκτή. Συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. χέρι δεκτή. 41 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή τελική ψηφοφορία άρκετη ψηφοφορία closed. Πέρας. Δεκτή. Συγχαρητήρια. Έκθεση Κοχμερίν. Ένα υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 σε 2 μέρη υπέρ του πρώτου κατά αποχές δεκτή δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 8 υπέρ κατά αποχές 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά να επαληθεύσουμε την 11 άρχεται η ψηφοφορία Πέρασε. Και απορρίπτεται. 12 υπέρ. Κατά. αποχές Δεκτή. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 19 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 22 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να επαληθεύσουμε την 22 άρχιτη ψηφοφορία. σφαίρας Απορρίπτεται. 24 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 25 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 26 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 27 υπέρ. Έχει αποσυρθεί. 28 υπέρ κατά εποχές δεκτή 29 υπέρ κατά εποχές δεκτή 30 υπέρ κατά εποχές να υπαλληθεύσουμε την 30 έρχεται η ψηφοφορία και πέρασε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 και βεβαίω συγκρίνεται. Και περνάμε στην εκτίση τη κυρίας ΕΚ. Είναι τελευταία. Να κάνουμε καμία επαλήθευση και ονομαστική ψηφοφορία. Συμβαστική 1. Ναι, υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 17 υπέρ κατά αποχές Συγκρίνεται. 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ κατά συγγνώμη. 32 Ευχαριστώ εδώ πέρα την Αντιπρόεδρο. 32 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβαστική 5 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβαστική 6 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 36 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. Συμβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 45 υπέρ, κατά, αποχέ, να επαληθεύσουμε. 45, να επαληθεύσουμε. Ε, άρχιτη ψηφοφορία, πέρας. Δεκτή. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 51 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβαστική 10 υπέρ. Κατά. Εποχέ. Δεκτή. Συμβαστική 59. Ξέχασα κάτι. Α, ναι. 58 υπέρ. Κατά. Εποχέ δεκτή. 59 υπέρ. Κατά. Εποχέ δεκτή. 60 υπέρ. Κατά. Εποχέ δεκτή. 62 υπέρ. Κατά αποχές 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 12 υπέρ πάλι που ξέφυγε 63 πρώτο μέρος ναι 63 πρώτο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτή Τώρα περνάμε στη 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 70 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 76. Πρέπει να τις ψηφίσουμε μία-μία ή μπορούμε να τις κάνουμε μπλοκ. Γίνεται. Όχι δεν γίνεται. 76 πέρα. Κατά. Αποχές δεκτή. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 79 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 80 υπέρ κατά αποχές δεκτή 81 υπέρ κατά αποχές δεκτή 82 υπέρ Α, η Λένα έκθελε το λόγο, παρακαλώ. Υπάρχει μια σύντομη προφορική τροπολογία της κυρίας Γκουτιέρης Ροντρίγκες. Θα ληφθεί υπόψη το κείμενο. Το θέμα της αγροδασονομίας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη όπως όλα τα θέματα της χρήσης γης σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και εγώ είμαι υπέρ αυτού. Τη δέχομαι λοιπόν αυτή την, την προφορική τροπολογία. Το δέχεστε με την προφορική τροπολογία. Λοιπόν, ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Παριθμόν 1. Αμπλόκ. Από 1 έως 9. Όλες τις λένε ΑΕΚ. Συμφωνείτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Σχεδόν ομόφωνα. Περνάμε λοιπόν στην τελική και τελευταία τελική ψηφοφορία. Τελευταία ψηφοφορία της ημέρας. Απολαύστε την. άρχη της ψηφοφορία. Πέρας. Και βεβαίω εγκρίνεται. Συγχαρητήρια. Να ευχαριστήσω τον συνάδελφο εδώ πέρα, ο οποίος κοίταγε και τον κατάλογο και χειρίζονταν και το μηχάνημα. Νομίζω θα πάρει ένα ειδικό βραβείο είτε των υπολογιστών είτε των γερμανών λογιστών. Λοιπόν, Ζητήσαμε όμως να μας μιλήσει η Κομισιόν για το σημείο 15. Οπότε, λίγη ισχύα, συνάδελφοι. Όσοι δεν θέλουν να ακούσουν, να περάσουν έξω ή να κάνουν ισχύα. Και σας παρακαλώ να μην, ξανακάνουμε, να μην ξανά τέτοιες ψηφοφορίες. Ε, ήταν, παρά ήταν. Κύριε Ρέμεκ, θέλετε να πείτε κάτι πριν ή να δώσουμε απευθείας το λόγο στην Κομισιόν. Ό,τι θέλετε. Μπορείτε να ρωτήσετε, να στραφείτε απευθεία στην Κομισιόν. Ωραία. Λοιπόν, ακούστε, αγαπητοί συνάδελφοι. Σας παρακαλώ, ήσυχα. Ε, Καρατήσαμε τον εκπρόσωπο της Κομισιόν ε, σε αναμονή ε, μέχρι τώρα. Λοιπόν, σας παρακαλώ. Κυρίες και κύριοι. Νομίζω ότι είναι σωστό να ε, προσέξουμε τη θέση της Επιτροπής. Η, η, η κυρία Κατερίνα Καβαδά. Ελπίζω να είπα σωστά το όνομά σας, κυρία Καβαδά. Απολύτως σωστά, ε, κύριε Πρόεδρε, ονομάζομαι Κατερίνη Καβαδά και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Ζητώ και εγώ συγγνώμη επειδή δεν ήρθα σήμερα το πρωί όταν ε, ε, ασχοληθήκατε εσείς με το ζήτημα. Στόχος αυτής της σύντομης παρέμβασή μου είναι να σας ενημερώσω για το την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργασίες ε, για την ενδιάμεση επισκόπηση των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής πλοήγησης. Όπως πολύ καλά γνωρίζετε, η Κομισιόν έχει και προγραμματική αλλά και νομική υποχρέωση να εμφανίζεται εντός ενώπιον του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με την έκθεση αυτή, επισημένοντας και ενημερώνοντάς σας ε, σε σχέση με το βαθμό ολοκλήρωσης και πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει πολλά πράγματα. Έχουμε να σας πούμε πολλά και για τις δυσκολίες και το τελευταίο διετή είχαμε αρκετές δυσκολίες. Να σας ενημερώσω επίσης και για τους κινδύνους που εμφανίστηκαν αλλά κυρίως για τις ε, μελλοντικές προκλήσεις και τις προοπτικές ε, σε σχέση με τον Γαλιλαίο. Ε, η... Κύριε Πρόεδρε, η Επιτροπή έχει γνωρίσει πολύ καλά ότι ε, ε, η Επιτροπή σας περιμένει την έκθεση τους τελευταίους 6-7 μήνες. Δηλαδή, από το Μάρτιο, ο κύριος Ρεμέκ, μετά από ε, περιμένει κάποια ένδειξη από πλευράς Κομισιόν για να μπορέσει να ε, τοποθετηθεί ενώπιον του Κοινοβουλίου σχετικά με τα, τις προκλήσεις και τα διάφορα θέματα του προγράμματος αυτού. Σήμερα λοιπόν θέλω να δικαιολογήσω ή τουλάχιστον να σας αιτιολογήσω την ε, καθυστέρηση αυτή. Τα αίτια είναι κυρίως τα εξής δύο που είναι συνδεδεμένα ε, και με θέματα προγραμματισμού αυτού του προγράμματος αλλά και με θεσμικά ζητήματα. Όσον αφορά τον προγραμματισμό, πρέπει να σας πω ότι η Κομισιόν ε, θα ήθελε μέσω της έκθεσης αυτής να ξεκινήσει μια σοβαρή και ουσιαστική συζήτηση με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και στο πλαίσιο αυτό η Κομισιόν θέλει να σας ε, επιδώσει ένα πλήρες, ε, ουσιαστικό και ρεαλιστικό έγγραφο. Και γι' αυτό περιμέναμε στοιχεία, κυρίως χρηματοοικονομικά, τα οποία θα είναι σταθερά και θα, μπορέσουν, θα μας έδιναν τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε σωστά την κατάσταση και να αναπτύξουμε ε, ρεαλιστικές προοπτικές. Σήμερα πλέον σας διαβεβαιώ ότι η Κομισιόν έχει αυτά τα χρηματοοικονομικά δεδομένα ε, δεδομένου ότι ολοκληρώθηκε αυτή η φάση ανάπτυξης και πρόκειται το 2011 να ε, σταλούν ε, αυτοί οι τέσσερις δορυφόροι. Έχουν ήδη ε, ε, υπογραφεί τέσσερις συμβάσεις το τελευταίο 25 Οκτωβρίου ενώ άλλες δύο αναμένονται στο τέλος του έτους ή στις αρχές του επομένου. Όσον αφορά τώρα το θεσμικό πλαίσιο. Παρότι το πρόγραμμα Galileo θέλει να προχωρήσει συνολικά ως ε, παροχή υπηρεσιών, πρέπει να ξέρουμε ότι ο, προ, ο κρηματοοικονομικός προγραμματισμός έπρεπε να, ε, συντονιστεί με το προγραμματισμό της Κομισιόν. Γνωρίζουμε ότι στις, 29 Οκτωβρίου, στις 19 Οκτωβρίου η Κομισιόν ενέκρινε μία ανακοίνωση για τον ε, κοινοτικό προϋπολογισμό και έκτοτε το πρόγραμμα Galileo, το πρόγραμμα Manager, δεν, ε, για αυτό το πρόγραμμα δεν υπάρχει παραμικρή αμφιβολία ότι δεν υπάρχουν πλέον επιπλέον ε, κονδύλια για το πρόγραμμα πριν από το 2014. Έχοντας λοιπόν στη διάθεσή μας όλα αυτά τα στοιχεία, η Κομισιόν, όπως ε, σας ανακοίνωσε την προηγούμενη φορά στο Στρασβούργο ο κύριος Ταγιάννη, η Κομισιόν λοιπόν σκοπεύει να προχωρήσει ε, σε, με βάση δύο φάσεις. Η πρώτη φάση που θα ξεκινήσει στο τέλος αυτού του χρόνου ή στις επόμενη, το, επόμενο έτος θα είναι η στις το επομενο ετος θα ειναι η εγκριση μιας ανακοίνωσης σχετικά με την πορεία του προγράμματος η οποία θα παρουσιαστεί στο Κοινοβούλιο αλλά και στο Συμβούλιο. Κύριε, ο κύριος Αντιπρόεδρος ε, περιμένει την επίσημη ανακοίνωση και σκοπεύει να ενημερώσει τα μέλη του Κοινοβουλίου αλλά και το Συμβούλιο ε, για τις βασικές ιδέες αυτού του εγγράφου που σκοπεύουμε να σας παρουσιάσω. Στη δεύτερη φάση, από τη στιγμή που θα κρίτησει με βάση αυτή την ανακοίνωση και επί τη βάση των κατευθύνσεων που θα προσδώσουν στην Κομισιόν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα προχωρήσουμε στο τέλος του 2011 υποβάλλοντας νομοθετικές προτάσεις για το Γαλιλαίο πάντα στο πλαίσιο των νέων χρηματοοικονομικών προοπτικών. Συνειδητοποιείται λοιπόν ότι για την Κομισιόν η εντατική συζήτηση που πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ ημών και ημών είναι εξαιρετικά σημαντική, ε, απολύτως απαραίτητη για την κανονική ε, ε, εξέλιξη του προγράμματος. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα εσείς και οι συναδελφοί σας να μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω επιθυμίζοντάς σας δύο πράγματα. Πρώτον, ότι τον Γαλιλαίο αποτελεί για την Κομισιόν, εξακολουθεί να αποτελεί, όπως και για σας, ένα στρατηγική σημασία πρόγραμμα. Ως ε, διαχειριστής του προγράμματος έχουμε την υποχρέωση, αλλά και την ε, δόξα να το δημιουργήσουμε όσο το δυνατόν ταχύτερα και υπό τις καλύτερες δυνατές συνθήκες ακόμα και χωρίς τα ε, επιπλέον κονδύλια μέχρι το 2014, στόχος μας είναι να διεισδύσουμε και να είμαστε έτοιμοι να διεισδύσουμε στην αγορά ήδη από το 2014 με τους 18 δορυφόρους που θα έχουν ήδη ε, σταλεί στο διάστημα ε, μέχρι τότε. Θα είναι σε θέση ο Γκαλιλαίο να δώσει και στους υπολίτες μας και στον κόσμο τρεις υπηρεσίες που, τις οποίες θα έχουν πρόσβαση ε, όλοι οι πολίτες μέσω πολλών εφαρμογών. Μέχρι σήμερα η Κομισιόν είχε τη χαρά να έχει τη στήριξη του Κοινοβουλίου. Ε, θεωρώ ότι... Ε, ε, έτσι θα συνεχίσει ε, να μας αντιμετωπίζει το Κοινοβούλιο, γιατί το πρόγραμμα αυτό δεν αποτελεί αποκλειστική πρωτοβουλία της Κομισιόν, αλλά μια κοινή πρωτοβουλία που όλοι καλούμαστε να στηρίξουμε. Είμαι στη διάθεσή σας για οποιασδήποτε, ε, να απαντήσω οποιασδήποτε ερωτήσεις. Παρατηρήσει εκτό μικροφώνου, δεν έχουν διερμηνήσει. Ναι, ναι, ήθελα να ευχαριστήσω λοιπόν την εκπρόσωπο της Επιτροπής για την πολύ σαφή της τοποθέτηση. Και όσον αφορά τη στήριξη του Κοινοβουλίου την οποία ζητά, θα ήθελα να, να υπενθυμίσω ότι μερικές εβδομάδες πριν έγινε μια μεγάλη ε, συνάντηση εδώ στο Κοινοβούλιο ε, που συνέπεσε με την υπογραφή του Γαλιλαίου ακριβώς ε, που καταδεικνύει τη σημασία που αποδίδει το Κοινοβούλιο στο Γαλιλαίο και ανοίγουμε τη συζήτηση. Ναι, ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι το πρόβλημα που έχουμε ε, με τον ε, Γαλιλαίο, ο κύριος Λαμπέρτς, ε, είναι ότι έχουν υπάρξει πολλές καθυστερήσεις. Είναι γεγονός ότι όλα αυτά τα δορυφορικά προγράμματα έχουν ξεπεράσει κατά πολύ το αρχικό τους κόστος. αλλά ακόμα ε, ε, έχουμε ήδη ξεκινήσει, έστω και αν δεν έχουμε φτάσει ε, σε κάποια αποτελέσματα, τουλάχιστον έχουμε ξεκινήσει. Αυτό που ακούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι μια ιδέα προγραμματισμού, μια ιδέα κόστους εφαρμογής του συνόλου του συστήματος ε, και δεν αναφέρομαι επομένω ε, στο υποσύστημα των 18 δορυφόρων αλλά στο πλήρε σύστημα των 24 ε, δορυφόρων και μας ενδιαφέρει να έχουμε ένα, ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα το οποίο θα λειτουργεί κανονικά Ξέρετε, δεν έχει έννοια το να δημιουργήσουμε ένα ενδιάμεσο πρόγραμμα 18 δορυφόρων. Θα πρέπει να δούμε επίσης και το κόστος ε, της μηδενικής επιλογής, δηλαδή της επιλογής του να σταματήσουμε. Τι θα γινόταν και ποιο θα ήταν το κόστος αν πάρουμε μια επιχειρηματική ας πούμε απόφαση λέγοντας ότι λαμβάνοντας υπόψη τις νέες εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αν σταματήσουμε ε, το κόστος θα είναι αυτό και αν συνεχίσουμε έτσι ώστε να ε, προσφέρουμε το ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το κόστος θα είναι αυτό γιατί αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια περιοχή που δεν είναι καθόλου ικανοποιητική. Από τη μία πλευρά δεν ξέρουμε αν θα έχουμε το σύστημα και αν θα λειτουργεί πλήρω. Ε, και εάν το σύστημα λοιπόν δεν λειτουργεί πλήρω, ε, τότε είναι ανώφελο. Δεν έχει έννοια να υπάρχει. Επομένω, εκεί ακριβώ είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το ερώτημα που πρέπει να απαντήσουμε και ακριβώ εκεί θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και τα χρήματά μα τα οποία δεν είναι και πάρα πολλά από ό,τι φαίνεται. Αυτό ήθελα να πω λοιπόν ότι ε, μέχρι ότου έχουμε έναν οικονομικό οδικό χάρτη πλήρη δεν μπορούμε να κάνουμε και πλήρη επιχειρηματολογία πάνω στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ πολύ Ράνστορφ. Ευχαριστώ. Ε, θα πω δύο λόγια μονάχα, γιατί προέρχομαι από χώρα η οποία ενδιαφέρεται πολύ για το πρόγραμμα Γαλιλαίο πρέπει να πω ότι είμαι εξαιρετικά απογοητευμένος από το μήνυμα που μόλις ελάβαμε. Σύμφωνα με το μήνυμα αυτό λοιπόν δεν ε, υπάρχει ε, καμία πρόοδος και επομένως καμία συγκεκριμένη ε, πληροφορία δεν μπορεί να συζητηθεί εδώ και επομένως εν κατακλείδη είμαι πολύ πολύ απογοητευμένος. Η κυρία Τικάου. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ την Επιτροπή για την παρουσίασή της. Θα ήθελα όμω να επιστήσω την προσοχή σα σε ένα σημείο και να κάνω και μία σύσταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αν μου επιτρέπετε. Δηλαδή, στο επόμενο πρόγραμμα ε, μέχρι το 2014 να δώσει επιπλέον χρηματοδότηση για την έρευνα. Γιατί όταν μιλάμε για τον Γαλιλαίο αναφερόμαστε βεβαίως στη δημιουργία μιας υποδομής. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι οι 18 δορυφόροι θα ξεκινήσουν, ναι, πολύ ωραία, αλλά αυτό δεν αρκεί. Ε, θα πρέπει να έχουμε πλήρη υποδομή και θα πρέπει να έχουμε και τις ε, υποδομές εδάφους θα πρέπει επίσης να έχουμε ε, και όλα τα αναπτυγμένα προγράμματα τα οποία θα μας επιτρέψουν να προχωρήσουμε και να ολοκληρώσουμε αυτές τις επενδύσεις. Μέχρι το 2018 γίνεται λόγος λοιπόν για τους 18 δορυφόρους και μετά θα ακολουθήσουν οι υπόλοιποι μέχρι το 2018. Περι... Εν όμως πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, να αναπτύξουμε τις υπηρεσίες και τις εφαρμογές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν τη στιγμή της ε, χρήσης ε, των δορυφόρων έτσι ώστε να έχουμε βέλτιστη χρήση των επενδύσεων που έγιναν για τον Γαλιλαίο. Η κυρία Χολ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι είναι εξαιρετικά μη ικανοποιητικό το γεγονός ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έχουν τόσο μικρή πληροφόρηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέχρι τώρα μας ζητούν μόνο να ψηφίσουμε για τα χρήματα και τους πόρους του Γαλιλαίου και αυτό δεν ε, μας ικανοποιεί. Θέλουμε να συμμετέχουμε και στις αποφάσεις, να έχουμε περισσότερη πληροφόρηση. Και νομίζω ότι θα συνεχίσω στην ίδια τροχιά των επικριτικών ε, σχολείων των συναδέλφων. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου ικανοποιητική αυτή η κατάσταση δεν μας δίδονται πληροφορίες ε, και πραγματικά δεν καταλαβαίνουμε αυτές τις καθυστερήσεις. Δεύτερον, η κυρία Τικάου και ο κύριος Λάμπερτς είπαν κάποια πράγματα. Εάν δούμε το κόστος πρέπει να έχουμε μια πλήρη αξιολόγηση ε, κόστους γιατί θέλουμε να ξέρουμε τι θα συμβεί εάν σταματήσει το όλο εγχείρημα. Από την άλλη πλευρά όμως με τρόπο διάφανο και ειλικρινή θα πρέπει να δούμε ποια είναι η επιστροφή που θα έχουμε, τι θα κερδίσουμε από ένα ήμι πρόγραμμα ή από την εφαρμογή ενός ενδιάμεσου προγράμματος. να ξέρουμε δηλαδή τι μπορεί να κάνει ο Γαλιλαίος, πόσο μπορεί να βοηθήσει τις ε, επιχειρήσεις, γιατί έχουμε βασιστεί πολύ ε, στο πρόγραμμα αυτό και νομίζω ότι είναι επικίνδυνα αυτά που μας ε, λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με ενδιάμεσες καταστάσεις, γιατί μέχρι τώρα μας έχει κοστίσει και πάρα πολύ χρήμα όλη αυτή η διαδικασία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Οντί. Εντυπωσιάζομαι κύριε Πρόεδρε η Κομισιόν έχει μια ευθύνη. Δεν απέδειξε παρά τα αυτά μέχρι στιγμής ότι είναι σε θέση να ε, δείξει ότι μπορεί να χειριστεί μεγάλα έργα. Εντυπωσιάζομαι από τους ε, συνοδέλφους εδώ, γιατί ήδη διαβάσαμε το ίδιο έγγραφο ή κάτι άλλο συμβαίνει. Ε, συζητήσαμε για τον Γαλιλαίο 100 ώρες. Ξέρουμε ότι είναι ε, ένα θέμα όπου τα έσοδα είναι μηδενικά. Βεβαίω τα επανέκτησε χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα κονδύλια. Όμω πρέπει διαρκώ να επενθυμίσουμε ότι πρόκειται ένα για ένα θέμα στρατιωτική ανεξαρτησία, υγεία και ασφάλεια που θέλει να κάνει η Ευρώπη. Δεν πρέπει να ε, εξαρτάται η Ευρώπη του Αμερικανούς. Αν ε, οι Αμερικανοί αύριο μας κόψουν ε, το σήμα ή αν έχουμε προβλήματα με την Κίνα, πρέπει να έχουμε τις δικές μας δυνατότητες. Πρέπει λοιπόν διαρκώς να μην αμφισβητούμε τις δυνατότητες. Το θέμα είναι εξαιρετικό από αυτούς τους υποδομής. Ας το υποστηρίξουμε. Πράγματι, συμφωνώ ότι πρέπει η Κομισιόν με μεγαλύτερες ταχύτητες και πιο ολοκληρωμένα να μας δίνει γραπτά τις ε, πληροφορίες. Συγκεντρώσατε το πάνελ Κοινοβουλίου-Συμβουλίου πολύ γρήγορα θεωρώ ότι πρέπει όλη η Επιτροπή, πέρα από το απλό πάνελ που θα συμμετέχουν 15-20 μέλη, ολόκληρη η Επιτροπή να ενημερωθεί για την κατάσταση προόδου αυτού του κεφαλαιόδου σημασία έργου ε, και που αφορά τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον κόσμο και αν ε, οι συνάδελφοι θέλουν να ξαναρχίσουν τη συζήτηση για το αν είναι πολιτικά σκόπιμο αυτό το έργο, πλέον θεωρώ ότι σε αυτή τη φάση όταν έχουν αρχίσει να εκτοξεύονται οι διάφοροι δορυφόροι, δεν μπορεί να συζητάμε για την σκοπιμότητα αν πρέπει ή όχι να γίνει το, το πρόγραμμα. Εγώ είμαι ικανοποιημένος από αυτά που μας ε, παρουσιάστηκαν, το χρηματοδοτικό, ε, η χρηματοδοτική πορεία και ανακοινώνεται ότι θα, γίνουν, ε, θα ληφθούν νομοθετικά μέτρα το 2011 σε σχέση και με τις διαπραγμα... οικονομικές διαπραγματεύσεις. Θεωρώ ότι έχουμε πρόβλημα. Γιατί αυτή η συζήτηση επαναλαμβάνεται διαρκώς. Μιλάμε για ένα έργο τεχνικής φύσεως. Δεν είναι κάποια δήλωση. Κάποιοι από εμά γνωρίζουμε ότι τα τεχνικά έργα έχουν διάφορες φάσεις. Παραδείγματος χάρη ημερομηνίε εκτόξευσης των δορυφόρων. Και είμαι βέβαιος ότι η Κομισιόν έχει κατά νου κάποιο χρονοδιάγραμμα μέχρι το 2013 και το 2014. Θα ήθελα όμως ξεκάθαρες ε, ευδιάκριτες πληροφορίες από την Κομισιόν για να ξέρουμε ποιες είναι οι σημαντικές φάσεις του προγράμματος. Πότε θα εκτοξευθούν οι 18 ε, δορυφόροι, τι είδους κάλυψη θα επιτευχθεί θα υπάρξει πλήρη κάλυψη, πλήρης κάλυψη, γιατί γι' αυτό από ό,τι γνωρίζω χρειάζονται 30 περίπου δορυφόροι. Θα ήθελα να ζητήσω τους φίλους της Κομισιόν να μας ενημερώσουν, να μας δώσουν αυτό το υλικό το ταχύτερο δυνατόν. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να καταλάβουμε ποιες είναι οι διάφορες ενδιάμεσες φάσεις και ποια είναι ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα και ποιο θα είναι το κόστος κάθε φάσης του έργου. Το έργο αυτό, τον Γαλιλαίο, είναι σημαντικό για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να θεωρούμε ότι δεν, ε, ε, είναι, ε, δεν βρίσκεται πλήρως υπό έλεγχο. Γνωρίζουμε τις τεχνικές δυσκολίες παγίδες, αλλά πρέπει να υπάρχει ένα είδος σχεδιασμού και προγραμματισμού, γιατί κάποιες τεχνικές προϋποθέσεις πρέπει να εκπληρώνονται. Πολλοί από εμά έχουμε ερωτήσεις για το τι εστί τον Γαλιλαίο, δηλαδή ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα. Και καλό θα είναι να πούμε ναι, μέχρι την τάδε ημερομηνία θα έχει ολοκληρωθεί το τάδε κομμάτι του προγράμματος, το, με την τη δίνα ημερομηνία άλλο κλπ. Δεν είναι σωστό να περιμένουμε μέχρι το 2013 ή το 2014. Υπάρχουν και άλλες εφαρμογές οι οποίες είναι εν αναμονή. Υπάρχουν δομές ε, ε, που, έχουν σχέση με την κοινή ωφέλεια και που εξαρτώνται από το αν θα τεθεί σε λειτουργία το σύστημα αυτό. Μέχρι στιγμής στηριζόμαστε στο αμερικανικό σύστημα GPS. Αν λοιπόν κάνουμε, ε, υπάρξει κάτι άλλο διαθέσιμο, κάτι που είναι καλύτερο, κάτι που προσθέτει περισσότερη αξία ε, στη, στους πόρους που, ε, διαθέτουμε. Ας γνωρίζουμε την κατάσταση και ποιος θα είναι ακριβώς ο στόχος που θα επιτευχθεί το 2012, το 2013 κλπ. Θεωρώ ότι και για την ίδια την Κομισιόν θα ήταν καλό κάτι τέτοιο θα πρέπει η Κομισιόν να γνωρίζει τι ακριβώς θα πρέπει να έχει γίνει το 2012, το 2013. Πρέπει το Κοινοβούλιο να ψηφίσει τα κονδύλια. Ιδάλλως θα καταλήξουμε εκεί που έλεγε ο κύριος Λομπέρ όσον αφορά τη δική μας Επιτροπή και όσον αφορά το σώμα, το Κοινοβούλιο, όσο λεπτομερέστερες είναι οι πληροφορίες, τόσο το καλύτερο. Θέλουμε να αποφύγουμε την ασάφεια και τα εδώ τις πληροφορίες που προέρχονται από δεξιά και αριστερά. Ξέρουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό το πρόγραμμα. Αυτό το Κοινοβούλιο πάντοτε στήριξε το πρόγραμμα Γκαλιλαίο και θέλει να λειτουργήσει το πρόγραμμα Γκαλιλαίο. Θα είναι τρομερό να διαλυθεί η στήριξη που έχει δώσει αυτό το σώμα και αυτό να οφείλεται στην έλλειψη πληροφοριών και στην ασάφεια. Εκτιμώ και το επαναλαμβάνω, εκτιμώ, καταλαβαίνω ότι είναι πρόγραμμα τεχνικό, δεν είναι θέμα δηλώσεων και αναγνωρίζουμε τα προβλήματα. Ευχαριστώ. Η κυρία Χόλ και πάλι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα να σχολιάσω αυτό το οποίο είπε ο κύριος Αούντι. Είπε είναι σημαντικό για την, ε, τον Γαλιλαίο είναι σημαντικό για την ε, στρατιωτική ανεξαρτησία. Όταν το Κοινοβούλιο ψήφισε υπέρ του Γκαλιλαίο, έγινε από πλευράς κομισιών σοβαρότατες αρνήσεις για τη ε, στρατιωτική διάσταση του προγράμματος. Μιλούσαμε για ένα πολιτική σημασίας ε, ε, πρόγραμμα με πολιτικές, πολιτικά αποτελέσματα. Τι έχει να πει η Κομισιόν όσον αφορά την σημασία του προγράμματος για τη στρατιωτική ανεξαρτησία παρακαλώ. Ο συνάδελφος κ. Λάμπερτ. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ με το ίδιο θέμα θέλω να ξεκινήσω. ίσως είμαι μια ειδική περίπτωση, αλλά και εγώ ε, δεν είμαι ε, αγαθός. Βεβαίως ε, είναι θέμα στρατιωτικής ανεξαρτησίας και βεβαίως έχει σημασία να έχει η Ευρώπη ένα ανεξάρτητο, ένα αυτόνομο ε, σύστημα ε, γεωγραφικής τοποθέτησης νομίζω ότι στον κόσμο που ζούμε δεν ε, ε, πρέπει να γνωρούμε κάποια πράγματα ότι ένα τέτοιο σύστημα έχει ε, στρατιωτικές σκοπιμότητες και συμφωνώ με αυτό. Τώρα το πρόβλημα που έχουμε είναι ότι βεβαίως μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στρατηγικά το χρειαζόμαστε. Αλλά πρώτον γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά όπως είπε και η Φιώνα ότι δεν θα έχουμε ένα μισό, ένα ε, μισό σύστημα δεν θα μας ικανοποιήσει. Δεν αμφισβητώ το ότι είναι χρήσιμο, αλλά το χρήσιμο θα είναι το ολοκληρωμένο σύστημα. Και έχουμε την εντύπωση ότι υπογράφουμε λευκές επιταγές. Μας λένε θα σας στοιχήσει τόσο και μετά διπλασιάζεται τριπλασιάζεται τετραπλασιάζεται το κόστος και δεν ξέρουμε που θα σταματήσει. Άρα το θέμα είναι να ξέρουμε τι, τι υπογράφουμε και για ποιο λόγο. Δηλαδή τι θα πάρουμε για τα χρήματα τα οποία δίνουμε. Και φυσικά εγώ πιστεύω στην αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον τομέα της άμυνας βεβαίως, αλλά όχι μόνο σε αυτό το τομέα, αλλά πρέπει να δούμε αν έχουμε τα μέσα για αυτή την αυτονομία και ε, μήπως φτάσουμε στα όρια μας με τα δημοσιονομικά και τι θα γίνει τελικά με αυτά τα χρήματα. Βεβαίως, ε, ε, ε ίσως μπαίνει το θέμα από το παράθυρο, αλλά σήμερα πρέπει να κάνουμε μια επιλογή, να πούμε θα πάμε υπέρ του πλήρους Γκαλιλαίου και αν μας κοστίσει μια καθυστέρηση, όχι όχι ε, ακύρωση 10 χρόνια καθυστέρηση, εντάξει. Αλλά εν τω μεταξύ να πούμε ποια θα είναι η επένδυση για να ξέρουμε τα χρήματα, τι πρέπει να δώσουμε. Όχι να μας λένε αυτό που δεν λέμε, να μας κάνουν να πούμε ότι θα το σκοτώσουμε τον Καλλιλέο, θα το εξαφανίσουμε κτλ. Όχι, δεν τίθεται. Όταν ξεκίνησε πριν από 10-15 χρόνια ήμουνα υπέρμαχος αυτής της ιδέας και λυπάμαι που χάθηκε ανάμεσα σε αυτά τα ΣΔΙΤ κτλ σαφώς πρόκειται για ένα έργο που το προωθεί το δημόσιο και η Ευρώπη. Και ξέφυγε σημαντικά, χρονικά και δημοσιονομικά και οικονομικά. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσουμε, να επανεξετάσουμε το νέο χρονοδιάγραμμα και τα νούμερα και να αποφασίσουμε. Εγώ δεν θέλω να αμφισβητούμε τις αποφάσεις μας κάθε τρία χρόνια, να πούμε μια συγκεκριμένη στιγμή. Αυτά έχουμε, υπογράφουμε και τελείωσε η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Για μία ακόμα φορά χαίρομαι που το Κοινοβούλιο θεωρεί τόσο σημαντικό θέμα τον ε, Γαλιλαίο και που δημιουργείται αυτή η συζήτηση, έστω και αν ε, τούτη τη στιγμή δεν έχετε τα στοιχεία τα οποία χρειάζεστε. Όλα αυτά τα ερωτήματα θα μας επιτρέψουν να επιβεβαιώσουμε κάποια στοιχεία και να αποσαφηνίσουμε κάποια άλλα. Θα ξεκινήσω αυτά τα οποία πρέπει να επιβεβαιώσω σήμερα. Δηλαδή ότι ο Γαλιλαίος δεν θα σταματήσει στους 18 ή στους 20 ή στους 24 δορυφόρους σου. Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συνόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι να υπάρξει το πλήρες σύστημα. Η Κομισιόν έχει κανονισμό, δηλαδή πρέπει να σεβαστεί ένα νόμο. Νόμο που ψήφισε και το Συμβούλιο και εσείς οι ίδιοι και που μας ζητά να έχουμε πλήρες σύστημα ικανό να παρέχει πέντε υπηρεσίες και βάσει αυτού του στόχου εργάζομαι και βάσει αυτού του στόχου ε, κάνω τον προγραμματισμό μου. Πέρα από, την, ε, από το στόχο όμως υπάρχει και η πραγματικότητα η οποία συνδέεται με τη χρηματοδότηση. Αυτή τη στιγμή με τα χρήματα τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας δεν είμαστε σε θέση να ξεκινήσουμε 28 ε, δορυφόρους. Άρα δύο δυνατότητες. Είτε σας λέω το αφήνουμε τελείως, είτε σας προτείνω τον τρόπο, την στρατηγική η οποία θα βελτιστοποιήσει την θέση σε ισχύ του συστήματος. Η στρατηγική που θα παρουσιάσει στην ανακοίνωση η Επιτροπή και μπορώ να σας το πω γιατί δεν είναι πλέον μυστικό, είναι να προχωρήσει σε φάσεις, σε καταστάδια. Ε, το πρώτο στάδιο θα είναι το 2014 με τις ε, open service, ανοιχτές υπηρεσίες, ε, την υπηρεσία Search and Rescue και την τρίτη υπηρεσία που θα είναι το PRS, Public Regulated Service. Γιατί, γιατί αυτό είναι ένα παράθυρο ευκαιρίας. Δεν μπορώ να περιμένω τους 28 ε, δορυφόρους για να ε, ρίξω το προϊόν στην αγορά. Θα πρέπει να δώσω στους ε, στους πολίτες την δυνατότητα να γνωρίσουν το Γαλιλαίο, να το μάθουν, να δουν ποιες είναι οι εφαρμογές του δεύτερο στάδιο από το 2016-2017 θα εξαρτηθεί βεβαίως ε, και από την χρηματοδότηση και πώς θα αξιολογηθούν ή, ε, συγγνώμη διορθώνει πώς θα εξελιχθούν οι συμβάσεις. Αλλά είναι στόχος ε, της Επιτροπής να μην κάνουμε συμβιβασμούς σε σχέση με τον αρχικό μας στόχο. Θέλω επίσης να σας πω ότι και εγώ δουλεύω 10 χρόνια το Γαλιλαίο Είμαι φανατική του Γαλιλαίου ε, και δεν είναι δυνατόν μετά από τόσα χρόνια να αρκεστούμε σε ένα ημισύστημα. Δεν υπάρχουν άλλωστε ημισυστήματα, υπάρχουν συστήματα. Ε, αυτό λοιπόν είναι ένα σύστημα το οποίο προχωράει αργά, αλλά το οποίο θα ολοκληρωθεί. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας ότι πριν αποφασίσετε επί της στρατηγικής θα πρέπει να έχετε στη διάθεσή σας όλα τα στοιχεία αυτή είναι μια εκ των ουκάνευ προϋπόθεση για την ε, Επιτροπή, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μέσω λοιπόν της ανακοίνωσής της σε δύο-τρεις μήνες ε, ήδη και πιο επίσημα μέσω μιας νομοθετικής ε, προτάσεως στα πλαίσια των νέων δημοσιονομικών προοπτικών η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως Program Manager και με την εμπειρία την οποία έχει θα είναι σε θέση να σας δώσει πληροφορίες πρώτον σχετικά με το πώς θα διαχειριστούμε το σύνολο του χρηματοδοτικού φακέλου που πριν από δύο χρόνια μας εμπιστεύτηκε το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, πόσα χρήματα έχουν ε, χρησιμοποιηθεί, ποιες ε, είναι ε, οι προσαυξήσεις και γιατί υπάρχουν οι προσαυξήσεις αυτές. Ε, σύμφωνα με την Επιτροπή, οι προσαυξήσεις αυτές δεν οφείλονται ε, σε κακή διαχείριση, αλλά τα άτομα τα οποία Όμως τα άτομα τα οποία καλούνται να συναποφασίσουν για το πρόγραμμα αυτό πρέπει να ξέρουν από τι προέρχονται ε, οι υπερκοστολογήσεις το πρόγραμμα αυτό επίσης θα πρέπει να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τους κινδύνους. Υπάρχει λοιπόν ε, τεχνική δυνατότητα ε, να, από το σχεδιασμό του δηλαδή ε, να γίνεται μία αναφορά, ένα reporting κάποιων δραστηριοτήτων, ναι, όχι. Και τέλος πρέπει να ξέρετε ποιο είναι το κόστος το κόστος, όχι ε, η μορφή χρηματοδότησης, ε, το κόστος της ολοκλήρωσης, γιατί στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δεν είναι να υπάρξουν 28 28 ε, ε, δορυφορικοί σταθμοί ε, σε τροχιά και κάποια επίγεια στοιχεία. Αλλά το στόχος της Επιτροπής είναι να εκμεταλλευτεί σωστά και επομένως να έχει καλά αποτελέσματα από αυτό το σύστημα. Γι' αυτό λοιπόν σε μερικούς μήνες θα σας υποβάλλω με μία πρώτη αξιολόγηση. Μία πρώτη εκτίμηση μέσα σε πολυετές πλαίσιο. Δεν θα κάνουμε αξιολόγηση η οποία θα είναι παγιωμένη σε 5 ή 10 χρόνια. Η εκμετάλλευση είναι κάτι που ξεπερνάει τους δημοσιονομικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι, ε, ε συνδέεται μάλλον στον προγραμματισμό ενός παγκοσμίου προγράμματος όπως είναι ο Γαλιλαίος και αν βρούμε κάποιον operator δεν θα, τον, δεν θα υπογράψουμε σύμβαση μαζί του για πέντε χρόνια ή για έξι. Θα πρέπει να έχει μια ιδιαίτερα ε, πολυετή έναν ιδιαίτερα πολυετή ορίζοντα. Σα ζητώ λοιπόν μερικέ εβδομάδε υπομονή έτσι ώστε να σα δώσουμε όλα τα στοιχεία τα οποία θα σα επιτρέψουν να προχωρήσετε σε καλύτερη αξιολόγηση τη ε, καταστάσεω και επομένω να είσαστε σε ε, καλύτερη θέση για να αποφασίσετε για το μέλλον του προγράμματος αυτού. Θα είμαι σύντομη, κύριε Πρόεδρε. Ε, αναφέρθηκε κάτι για τον ρόλο και την χρήση των προγραμμάτων έρευνας. Ο Γαλιλαίος βεβαίως γνωρίζει τις ε, ευκαιρίες αυτές. Μέχρι τώρα έχουμε τη στρατηγική να πληρώνουμε ε, το, την υποδομή του Γαλιλαίου μέσα από την δική του γραμμή του προϋπολογισμού, αλλά μπαίνοντας ε, στην δημιουργική σφαίρα της αγοράς, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα, τα χρηματοδοτικά μέσα για τα προγράμματα και βάσει αυτού του στόχου θα συνεχίσουμε και στα επόμενα έτη. Ολοκληρώνω λέγοντας ότι ο αρμόδιος επίτροπος και οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται πάντα και θα βρίσκονται στη διάθεσή σας για να συζητήσουν οποιοδήποτε σκέλος του προγράμματος, για να συζητήσουν οποιοδήποτε θέμα συνδέεται με το πρόγραμμα αυτό. Μπορείτε απλώς να μας υποβάλλετε ένα αίτημα, θα είμαστε πάντα στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σοντή, θέλει να κάνει μια παρατήρηση ακόμα, όχι. Ωραία. Οπότε σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα οποία μας είπατε. Ναι, παρακαλώ, συγγνώμη. I'm sure it was but you didn't actually ε, φαντάζομαι πως κατά λάθο έγινε, αλλά δεν απαντήσετε το ερώτημά μου για την ε, στρατιωτική ανεξαρτησία. Έχετε δίκιο, ζητώ συγγνώμη μεταξύ των σημείων που θέλω να επαναβεβαιώσω είναι ότι ο Γαλιλαίος είναι ένα ε, μη στρατιωτικό ε, πρόγραμμα ε, που ελέγχεται από μη στρατιωτικούς φορείς. Όμως μεταξύ των πιθανών εφαρμογών θα μπορούσε να θα μπορούσαν να υπάρξουν εφαρμογές κρατικές και ενδεχομένως και στρατιωτικές. Όμως δεν θα πρέπει να συγχαίωμε μεταξύ εν, της ύπαρξης ενός στρατιωτικού συστήματος ή της ύπαρξης ενός συστήματος που θα μπορούσε να εφαρμοστεί ε, και στον στρατιωτικό τομέα. Η διαφορά είναι τεράστια. Επίσης, πριν από ένα μήνα, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο εκλήθησαν να εργαστούν επί προτάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τις αρχές πρόσβασης των χρηστών ε, στις υπηρεσίες ε, PRS. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει συζητήσεις ε, στο Συμβούλιο μπορούμε να συζητήσουμε την ίδια πρόταση και στο Κοινοβούλιο, γιατί έτσι κι αλλιώ η πρόταση θα πρέπει, η, συγγνώμη, η απόφαση θα πρέπει να ληφθεί από το Συμβούλιο αλλά και από το Κοινοβούλιο. Ε, είμαστε στη διάθεσή σα λοιπόν να ρίξουμε όσο φω χρειάζεται ε, σε αυτά τα θέματα. Επίση, τον μήνα Ιούλιο ε, υπήρξε η έκθεση τη κυρία Κόπα, η οποία έλαμβανε υπόψη τη τα στοιχεία αυτά και η οποία διαφοροποίησε το Civil System Under Civil Control, μη στρατιωτικό σύστημα το οποίο θα ελέγχεται από μη στρατιωτικούς φορείς και ε, σύστημα το οποίο μπορεί να έχει και στρατιωτική εφαρμογή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σας πω πως ήταν η πρώτη φορά που παρουσίασε η Κομισιόν τα πράγματα λογικά και κατανοητά για μένα τουλάχιστον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας βοήθησε αυτό και Σα παρακαλώ να ακούσετε αυτά τα οποία είπαν οι συνάδελφοι. Καλό είναι να λαμβάνουμε πάντα τα νέα δεδομένα έστω και σε ένα έγγραφο γιατί δεν είναι όλοι οι συνάδελφοι εδώ πέρα πάντα οπότε μπορούμε να τα διαβάσουμε και δεν χρειάζεται να είναι πολύ σελίδο, μία-δύο σελίδες με μία σύντομη είδηση, μία παρατήρηση. Θα μα βοηθήσουν πάρα πολύ στον περαιτέρω μας. κύριος Ρέμεκ. Předsedo, já bych jenom chtěl poděkovat eh, všem kolegům a kolegyním za eh, aktivní přístup a za jejich připomínky. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα απλώ να ευχαριστήσω όλους όσοι συνεισέφεραν ε, στη δουλειά μου και όλοι όσοι συνεργάστηκαν, όλους όσοι συνεργάστηκαν μαζί μου. Θέλω να ευχαριστήσω την Κομισιόν για, και την εκπρόσωπό της για την ε, βοήθεια και τη συνεισφορά. Δεν πιστεύω ότι χρειάζεται να αλλάξουμε το παραμικρό σε αυτά που σήμερα το πρωί αποφασίσαμε. Οι συνάδελφοι πραγματικά στήριξαν την άποψή μου ότι δηλαδή δεν έχουμε επαρκή γνώση και πληροφορίες και έκανα και κάποιες προτάσεις για το τι μπορεί να γίνει. Όλα αυτά ισχύουν πιστεύω και αξίζει να συντάξω μια επιστολή με βάση αυτά που συμφωνήσαμε σήμερα το πρωί. Τώρα όσον αφορά το θέμα της, του να κάνουμε μια έκθεση έστω και ανεπίσημη για τα θέματα δορυφορικής ε, πλοήγησης Θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή η πολιτική του διαστήματος, συμπεριλαμβανομένου και του Γαλιλαίου, ε, χρειάζεται μια πολύ πιο πολιτική προσέγγιση. Μέχρι ότου συνειδητοποιήσουμε και καταφέρουμε να γίνει αντιληπτό ότι πρόκειται αυτό εδώ για ένα έργο υποδομής, το οποίο επηρεάζει όλες τις πολιτικές και όλους τους τομείς της ζωής μας, δεν θα καταφέρουμε να εξηγήσουμε το λόγο για αυτό το κόστος. Το έχουν πει και άλλοι συνάδελφοι, αυτό το λέω, το επαναλαμβάνω για, λόγους, για να είμαι ολοκληρωμένο. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που έγινε στη Βρετανία, η δραστηριότητα που αφορά το διάστημα ε, ε, δεν ε, υπόκειται στους νόμους της ύφεση. Δηλαδή, αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο κινείται στο επίπεδο των 7,5 δις ε, λιρών και αυξάνεται τα τελευταία χρόνια διαρκώς. Ε, αυτές είναι οι πληροφορίες που έχω λάβει. Δηλαδή ένα σύστημα δορυφορικής πλοήγησης δεν θα μας είναι καθόλου χρήσιμο αν προχωρήσουμε όπως πάμε τώρα. Δηλαδή αν το προσεγγίσουμε ε, με μια μέθοδο σαλαμοποίησης στην ουσία αυτό θα σήμαινε σαν να φτιάχνουμε, ας πούμε ένα σιδηροδρόμο και βάζουμε μόνο τη μία ράγα. Αυτό περίπου κάνουμε, προσπαθούμε να κάνουμε με τον Καλλιλέο. Άρα ολοκληρώνοντας θέλω να πω ότι πρόκειται για την πρώτη φορά που η Ευρώπη κατάφερε να έχει στη διάθεσή της ένα εγγυημένο πολιτικό έργο κανένας από τους άλλους οι οποίοι προσέφεραν τέτοιο σύστημα δεν εγγυώνται τις πολιτικές υπηρεσίες. Δεν θεωρώ ότι μπορεί κανείς να πει ότι η Ευρώπη δεν έχει την οικονομική ισχύ να κάνει αυτό το οποίο κάνει η Ρωσία ή η Αμερική. Πρέπει πιστεύω να είμαστε σε θέση να βρούμε τα κεφάλαια που αντιστοιχούν στο έργο που θα αποδώσει αυτό το πρόγραμμα. Όλοι πιστεύω μιλήσανε και περί, λίγο πολύ συμφωνούν. Ε, η έκθεσή μου αυτό μπορεί να το διατυπώσει ώστε να στηριχθεί το πρόγραμμα αυτό με την πολιτική υποστήριξη που του αξίζει. Ωραία, σας ευχαριστώ. Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω την ε, Κομισιόν να μας ενημερώνει. Αυτά σας ευχαριστώ και εύχομαι καλό διάλειμμα.